Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε με το σημείο 10 της ημέρησης διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μάικλ Σνάιντερ, που είναι ο εισηγητής της αγρομοδότησης ε, της Επιτροπής των Περιφερειών για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Στην ομάδα εργασία για το μέλλον της πολιτικής συνοχή είχαμε ήδη ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Σνάιντερ και εκφράσαμε όλη την επιθυμία στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να ακούσουμε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Χωρίς άλλη χρονοτριβή λοιπόν, σου δίνω το λόγο Μάικλ. Ευχαριστώ πολύ Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ κυρία Χιούμπνερ για την πρόσκληση. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συμμετέχω σε εργασίες της Επιτροπής σας. Θα πρέπει να επισημάνω βέβαια ότι για εισηγητή της Επιτροπής των Περιφερειών έχει μεγάλη σημασία το να μπορώ να έρχομαι εδώ, να μιλάω μαζί σας, να παρίσταμε στις ε, διαβουλεύσει, συζητήσει, σα να ακούω απόψεις και στις δικές, τις μου. Είναι αυτό που λέμε και οι δύο κερδίζουν. Ε, έχουμε να κάνουμε δηλαδή, εν προκειμένου, με μια προοπτική γνωμοδότηση, όπως την ονομάζουμε, perspective, ε, δηλαδή συζητούμε τι μπορούμε να προτείνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική συνοχής και θέλουμε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο ετοιμάσαμε αυτόν τον Απρίλιο εφέτος, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και στις 15 Απριλίου του 2010 υιοθετήθηκε η γνωμοδότηση. Με χαρά μπορώ να σας πω ότι εγκρίθηκε ομόφωνα Ε, βέβαια, εύκολο ίσως το που θα μου πείτε είναι να γράψει κανείς ε, γνωμοδότηση συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επιθυμίες και μην βάζοντας τίποτα που να ενοχλεί τον ένα ή τον άλλον. Αλλά δεν συνέβη έτσι. Ήταν μια γνωμοδότηση στην οποία δουλέψαμε πολύ και η οποία όντως ικανοποίησε τις ε, απαιτήσει της πολιτικής συνοχής και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε μια καλή θέση εκ μέρου τη Επιτροπή των Περιφερειών για την Πολιτική Συνοχή. Κυρίε και κύριοι, δεν θέλω να σα κάνω παρουσίαση τεχνοκρατικού τύπου σήμερα. Τι ε, λεπτομέρειε πολύ ευχαρίστω εάν θέλετε να εμβαθύνουμε. Είμαι στη διάθεσή σα. Θα κοιτάξω όμω περισσότερο τι μεγάλε γραμμές της πολιτικής που προτείνουμε εμείς, κάνοντας παράλληλα και μια αναφορά, μια επισκόπηση στην φυστάμενη κατάσταση. Η κύρια τοποθέτηση λοιπόν, την οποία διατυπώνουμε σε σχέση με τη γνωμοδότηση αυτή για τη μελλοντική πολιτική, είναι ότι στηρίζουμε την συνέχιση ισχυρής και αηφόρου πολιτικής συνοχής, πολιτικής συνοχής που επίσης θα έχει κάτι να προσφέρει σε κάθε περιφερειακή η τοπική αρχή. Μας καθοδηγεί η πεποίθηση πως η πολιτική συνοχής, όπως καμιά άλλη στην Ευρώπη, καμιά άλλη ευρωπαϊκή πολιτική, μπορεί να προσφέρει για τον κάθε πολίτη ορατή πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτική που καθιστά στον πολίτη ορατή την Ευρωπαϊκή Ένωση και απτή και τον βοηθάει μέσα από τις διαδικασίες τις κοινωνικές και τις οικονομικές στην Ευρώπη. Και έτσι και σήμερα επισημαίνουμε πόσο στο μέλλον και το διατυπώνουμε αυτό μέσα στην έκθεση, θα πρέπει να διατηρήσει η πολιτική συνοχή σημαντικό τμήμα των κοινοτικών κονδυλίων για τις δραστηριότητες της σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών. Βέβαια, τα θέματα τα δημοσιονομικά δεν τα συζητούμε μόνο σε αυτό το πλαίσιο, αλλά σε αυτή την γενική τοποθέτηση μόνο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κύριες ε, απαιτήσει που διατυπώσαμε από το έγγραφο. Επίσης, συμμεριζόμαστε τις απόψεις Επιτροπής ε, εν της ε, κοινωνικής και οικονομικής εδαφικής συνεργασίας και συνοχής να έχουμε ιδιαίτερη έμφαση στις κλιματικές αλλαγές, ε, τις δημογραφικές εξελίξεις, την παγκοσμιοποίηση, την προστασία του περιβάλλοντος. Όσο δεν αφορά την πολιτική συνοχής, εκφράζουμε την πεποίθησή μας πως οι νέες προκλήσεις είναι και προκλήσεις για την πολιτική συνοχή. Είναι προκλήσεις για την πολιτική συνοχή εφόσον θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε ε, για να συμβάλλουμε μάλλον στην ε, αντιμετώπιση των ε, οικονομικών και κοινωνικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προβλήματα αυτά δηλαδή μπορεί η Ευρώπη καλύτερα να τα αντιμετωπίσει με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών της. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν σημειώνεται ανάγκη για ριζική αλλαγή των βασικών διεθνωτικών μέσων ή για προσθήκη νέων στόχων, συγκεκριμένων στοχεύσεων μέσα στην πολιτική συνοχή. Κυρίε και κύριοι, στη γραμμοδότησή μας υπογραμμίζουμε και το επισημαίνω αυτό έχοντας και τα μάτια στραμμένα στην, ε, έχοντας υπόψη την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που μας έχει πλήξει εδώ και δύο χρόνια, πώς η, οικονομική, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής σύνοχης, της συνύπαρξης της κοινωνικής, αλλά και στην μείωση των κοινωνικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με δεδομένη την κρίση, ακριβώς θα πρέπει η πολιτική επιλογή της διαμόρφωσης της κοινωνικής ε, συνοχής να αποτελέσει ένα όλο μαζί με την οικονομική και την εδαφική συνοχή και να μην παραμεληθεί μετά το πέρας της περίοδου, δηλαδή μετά το 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤΑΦ, μπορεί να αποτελέσει το πιο σημαντικό όργανο για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, για την επιτεύξη των στόχων αυτών και στο μέλλον. Και ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να διατηρηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να αποτελέσει μέσω ολοκληρωμένης επέμβασης μαζί με όλα τα άλλα μέσα που προβλέπονται για την πολιτική συνοχή. Ιδιαίτερα στην γνωμοδότησή μας δε καταγράφουμε την βασική ε, πεποίθησή μας ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία ότι αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο, πολύ σημαντικό μέσο και το σημαντικότερο, ώστε όλες, όλες υπογραμμίζουν οι περιφέρειες να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη της ενδογενούς τους, του ενδογενούς τους δυναμικού ε, και αυτό με μία αισιόδοξη θα έλεγα θεώρηση την οποία μπορώ να πω ότι αρχίσαμε να διαπιστώνουμε ήδη όταν είχαμε επίτροπο την κυρία Χιούμπνερ την θετική δηλαδή θεώρηση του γεγονότος ότι κάθε περιφέρεια έχει ένα δυναμικό, έχει δυνατότητες και δυναμικό ανάπτυξης, εξέλιξης, δυναμικό το οποίο πρέπει κανείς να αφυπνήσει, να αναπτύξει, να αξιοποιήσει. Και γι' αυτό η κύρια μας ε, πεποίθηση εδώ, που εκφράζουμε εδώ, είναι ότι το Ταμείο Συνοχής δεν είναι απλώς δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα είδος φιλανθρωπικής πολιτικής. Δεν είναι ελεημοσύνη προς ε, ζητιάνους. Είναι μία ουσιαστική επένδυση για το δυναμικό που υπάρχει, που μπορεί να αναπτυχθεί, που πρέπει να αναπτυχθεί μέσω ή μακροπρόθεσμα στις περιφέρειες αυτές, μπορεί να τις βοηθήσει να εγκαταστούν αυτόνομες και αυτοδύναμες. Και αναφερόμενος και σε κάποιες από τις παρατηρήσεις του Φεντερίκο Μπάκα μέσα στην δική του έκθεση, ευελιξία και ε, πρόσδοση δυνατοτήτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και την, ε, το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ελευθερίας επιλογής για τις περιφέρειές μας, για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και έτσι και με την πρόσδοση βέβαια, με τον προσδορισμό των προϋποθέσεων, αλλά και ταυτόχρονα την ύψιστη δυνατή ευελιξία μπορούμε να εξυπηρετήσουμε παραπέμποντας φυσικά και στην αρχή της επικουρικότητας, αυτό το καταγράφουμε ξεκάθαρα στην χρωμοδότησή μας, μπορούμε λοιπόν να παραπέμψουμε στην αρχή της επικουρικότητας και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής καταγράφουμε κάποιες βασικές αρχές με βάση τις οποίες εργαζόμαστε, επιγραμματικά θα σας τις αναφέρω. Οι αρχές λοιπόν, μερικές από τις αρχές μας είναι και για το μέλλον διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής με βάση στόχους για ολόκληρη ε, στόχους που να μην είναι γενικοί, γενικόλογοι όλων, ε, για όλη την Ευρώπη, δηλαδή θα έλεγα επανεθνικοποίηση των στόχων, ιδιαίτερη στόχευση στις περιοχές που έχουν ε, ανάγκη, προσφορά όμως για κάθε περιφέρεια, διατήρηση δηλαδή της προσφοράς των δυνατοτήτων για κάθε περιφέρεια και διατήρηση της αποκεντρωμένης προσέγγισης και ταυτόχρονα είμαστε πεπισμένοι ότι για την πολιτική συνοχής η προσέγγιση στα, στην κυκλική δομή των ε, ταμείων είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και στο μέλλον. Το λέω αυτό ε, εντό παρενθέσεως γιατί έχω ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη δική μου την περιφέρεια αλλά και ε, σε άλλες περιφέρειες το έχουμε διαπιστώσει. Εγώ από το Σάξεν, από τη Σαξονία δηλαδή, Σαξενάνχαλτ, βλέπω ότι εμφανίζεται ένα πρόβλημα το οποίο και εσείς έχετε επισημάνει και σε αυτή τη χρονική περίοδο, την λειτουργική μάλλον περίοδο, ε, χρησιμοποιούνται κονδύλια, ναι, πλην όμως έρχεται μετά το ελεγκτικό συνέδριο και απαιτεί την ε, διαπίστωση της χρήσης αυτών των κυκλικών ε, κονδυλίων σε συγκεκριμένους στόχους, φερρυπίν κλιματική αλλαγή κτλ. Και μετά ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση από το, ταμείο, από το Ελεκτικό Συνέδριο, το Ταμείο Συνοχής, την Επιτροπή των Περιφερειών, τη δική μας την Περιφέρεια, για να δούμε πώς μπορούμε να αποδείξουμε και μάλιστα μερικές φορές εάν είναι πιο ε, ευρύς ε, ο στόχος θα πρέπει να Ε, θα πρέπει να τον περιορίσουμε έτσι ώστε, ίσω όχι κατά γραφειοκρατικό τρόπο, αλλά πάντω να στοχεύει καλύτερα του στόχου οποίου απαιτεί το ελεκτικό συνέδριο. Για τη μελλοντική αρχιτεκτονική τη πολιτική συνοχή, πάλι μπορώ να σα πω σύντομα δύο λόγια, είναι οι θέσει οποίε και εσεί έχετε ε, υποστηρίξει. Δηλαδή, στο μέλλον θέλουμε η πολιτική οι περιφέρειες εκείνες οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί με τους ίδιους ρυθμούς, δηλαδή οι πιο μειονεκτούσες, να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των μέσων ε, των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Επίσης, επί μακρόν συζητήσαμε το ζήτημα της ε, ε, διάκρισης, των, της οριοθέτησης των περιφερειών. Με ποιους δείκτες οριοθετούμε τις περιφέρειες και πρέπει να σας πω ότι από τη δική μας συζήτηση στην Επιτροπή των Περιφερειών είναι σαφές πως το ΑΕΠ μπορεί να αποτελέσει έναν δίκτυ αξιολόγησης και διάκρισης των ε, ε, περιφερειών που έχουν μεγαλύτερη και λιγότερη, ανάπτυξη και θα πρέπει να διατηρηθεί ως κριτήριο. Υπάρχουν και άλλα επίπεδα στα οποία μπορούμε να ορίσουμε δείκτες, όπως παραδείγματι αξιολόγηση των επιτυχιών της πολιτικής συνοχής, όπου πρέπει να δούμε αν θέλουμε να έχουμε περισσότερους και καλύτερους δείκτες, αλλά πάντως όχι ε, ως κριτήρια για την οριοθέτηση για το χαρακτηρισμό των περιφερειών. Επίσης, σε σχέση με τις περιφέρειες που βλέπουμε να βγαίνουν από, την, ε, από τους στόχους το 2013, μεταβατικές λεγόμενες περιφέρειες, θέλουμε εκείνες οι οποίες έχουν ξεπεράσει προς τα άνω το όριο του 75% για την προσεχή περίοδο, να διατηρήσουν την στήριξη κατά όρους πιο ε, γενναιόδουρους, περισσότερη δηλαδή στήριξη θέλουμε από ό,τι προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν επενδυθεί επιτυχημένα και ακριβώς αυτές τις σοβαρότατες επενδύσεις, σημαντικότητες επενδύσεις θέλουμε να διατηρηθούν, θέλουμε να καταστούν αηφόρες και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να μειωθούν ριζικά τα κονδύλια στις περιφέρειες αυτές γιατί θα προκαλούσε κάτι τέτοιο μεγάλο πλήγμα ω προς την αηφορία και τη διαφύλαξη των στόχων που επιδιώχθηκαν με αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Και επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει και στο μέλλον η εδαφική συνεργασία να ενισχυθεί η υπερσυνοριακή, η διασυνοριακή και η περιφερειακή συνεργασία. Η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία προσθέτει και αυτή από πλευράς της η συνεργασία και η συνύπαρξη των περιφερειών μπορεί να αποτελέσει πιστεύω ένα ε, ιδιαίτερο στόχο. Ως προς την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής, θα ήθελα να πω δύο λόγια γενικά. Φυσικά, κατάργηση της γραφειοκρατίας, ε, των περικών, περί των γραφειοκρατικών ε, ε, ρυθμίσεων κτλ. είναι στόχοι. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε περισσότερη ευελιξία με το βλέμμα στραμμένο προ τι ιδιαιτερότητε τη εθνικές, αυτό το βλέπουμε ήδη και κατά την υλοποίηση αλλά και κατά τον έλεγχο τη διάθεση των κονδυλίων, ότι δεν υπάρχει επαρκή εξέταση, λήψη υπόψη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και γι' αυτό καλύτερο θα ήταν και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, συνέδρια να συμμετέχουν στη διαδικασία του ελέγχου του τρόπου με τον οποίο διατέθηκαν τα ε, κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Και προχωρώ προς ένα τελευταίο σημείο, κυρίες και κύριοι, για να περιοριστώ περισσότερο και την ομιλία μου στον χρόνο που με έχει διατεθεί, ως προς την στρατηγική Ευρώπη 2020 και την αναφορά στην διαρθρωτική πολιτική. Η Επιτροπή των Περιφερειών, τόσο στην γνωμοδότηση αλλά και πέραν αυτής ε, στην ανάπτυξη, έχουμε συμμετάσχει στην ανάπτυξη στρατηγικής του, της Ευρώπης 2020. Ήταν μια πρώτη πρόταση που ξεκίνησε χωρίς καν την αναφορά της πολιτικής συνοχής, χωρίς αναφορά στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στη συμμετοχή της ενδιαφικής διάστασης, στην αρχική πρόταση. Βελτιώθηκε σημαντικά με την πρόταση της Επιτροπής το Φεβρουάριο, ε, τουλάχιστον στα λόγια, στο γράμμα, αναφερόταν ε, η πολιτική συνοχή, η εδαφική συνοχή κτλ. Αλλά πέραν αυτών των ανακοινώσεων της Επιτροπής νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση των προτάσεων ως προς το εξής και πάλι επιγραμματικά θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ότι δεν είναι δυνατόν η πολιτική συνοχή στο μέλλον να αποτελεί ένα απλό μέσον εφαρμογής μιας προσωρινής στρατηγικής της Ευρώπης του 2020 δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτό το ρόλο μόνο. Κύριες πρωτοβουλίες λοιπόν που προτείνονται μέσω από αυτήν τη στρατηγική δεν μπορούν να περιορίζουν το πεδίο δράσεως της πολιτικής συνοχής για τα διευθυντικά ταμεία ε, έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα τα επίπεδα στο τοπικό, το περιφερειακό επίπεδο και αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση και επίλυση προβλημάτων δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω του περιορισμού των, ε, της πρικοδοτήσεως ε, και των συγκεκριμένων τομεακών καθηκόντων ή εντολών που προσδίδονται στην πολιτική συνοχή. Έτσι λοιπόν θα ήταν πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι έχει χάσει την σημασία του μέσα σε αυτή τη στρατηγική του 2020 η ε, αρχή της επικουρικότητας έχει σχεδόν λησμονηθεί. Δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά στην, όπως είχαμε με τη στρατηγική της Λισαβόνας, στις τοπικές περιφερειακές αρχές στην επικουρικότητα. Και αν πούμε ότι απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας, αυτό ασφαλώς οφείλεται στο ότι δεν ήταν καν επαρκής από εκείνη την εποχή ήδη η προβολή των τοπικών, των περιφερειακών αρχών και η ανάδειξη των δυνατοτήτων τους για ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα για το, το οποίο θα πρέπει να μας καθοδηγήσει στο μέλλον και το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο να συνυπάρξουν κατά τρόπον οργανωμένο και εδώ κλείνω, ε, ε, υποδεικνύοντας ε, κυρίες και κύριοι ότι με τον κύριο Λάμπερτ Φωνίσλ Ρόι, τον κύριο συνάδελφο, έχουμε συζητήσει το πώς θα μπορούσαμε όλες αυτές τις ιδέες και ανησυχίες να τις εγγράψουμε μέσα σε ένα σύμφωνο, σύμφωνο εδαφικής συνοχής. Ήδη σήμερα ε, δημοσιεύθηκε η δήλωσή μας, την οποία, ξέρω θα λάβετε γνώση όλοι και ελπίζω ότι θα μπορέσετε και εσείς να συμφωνήσετε και να ακολουθήσετε αυτή την πρωτοβουλία. Την προσεχή εβδομάδα θα έχουμε να συζητήσουμε στην Επιτροπή των Περιφερειών ένα ψήφισμα αντίστοιχο, δηλαδή το ψήφισμα το σχετικό με την πρόταση για ένα ε, σύμφωνο εδαφικής συνοχής, ένα εδαφικό σύμφωνο. Αυτά είχα να πω κυρίες και κύριοι, ως κύρια στοιχεία της ε, έκθεσής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σνάιντερ, τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Νιστερόη πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, είναι καλό που έχουμε ξεκινήσει νωρίς τη συζήτηση για να ενημερωθούμε. Ποια είναι η άποψη των τρίτων. Εμείς Δεν έχουμε όλες τις απόψεις εδώ όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Ξεκινήσαμε φέτος. Καλό θα ήταν να δουλέψουμε με ομάδες εργασίας. Ορισμένοι έχουμε προσκληθεί, είναι αλήθεια, που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα λοιπόν έχουμε βάλει κάποιους θεμελιώδεις λίθους. Από εδώ και πέρα πρέπει να χτίσουμε το οικοδόμημα αυτό της πολιτικής συνοχής για το μέλλον. Συνεπώς, πρέπει ως Επιτροπή Περιφερειών να δούμε εμείς τι θέλουμε και να συζητήσουμε εμείς ώστε να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Συγχαρητήρια πάντως για αυτά που άκουσα, τα διάβασα και όλα. Όντως είναι κάτι που καλύπτει το όλο είναι και η Επιτροπή των Περιφερειών που συμμετέχει. Το είδα αυτό το έγγραφο. Και τώρα καταλαβαίνω ότι ομόφωνα υπάρχει αυτό το The Driving Force που έχει ετοιμαστεί, αλλά μάλλον εδώ πέρα εκπροσωπεί το ολόκληρη Επιτροπή των Περιφερειών. δεν ε, ξεκινάτε με την αναδιάταξη της αρχής ε, της συνοχής. Εσείς αναφέρεστε στις μεθόδους με τις οποίες έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα για τη συνοχή. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι σε επίπεδο Ευρώπης και ΑΕΠ κατά κεφαλή, ότι αυτά είναι τα κυριότερα κριτήρια τα οποία θέλουμε να κρατήσουμε. Το ΕΛΚ το στηρίζει αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει βέβαια να δούμε και την εδαφική διάσταση στα κράτη-μέλη, έτσι όπως έχουν τα λειτουργικά προγράμματα, αλλά να προσπαθήσουμε κάπως σε λεπτομέρειες, σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο να αναλύσουμε την κατάσταση. Τώρα βέβαια έχουμε την κρίση. Δεν ξέρουμε καλά-καλά όταν εμείς θα καθορίσουμε τα κριτήρια, ποιες περιφέρειες θα ανήκουν σε ποια κατηγορία. Πώς θα έχει διαμορφωθεί η Ευρώπη τότε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί οι περιφέρειες ε, ορισμένες σήμερα μπορεί να είναι μια χαρά και μετά από ένα χρόνο τα νέα στοιχεία που θα έχουμε να είναι εντελώ διαφορετικά. Όταν υπάρχουν περιφέρειες με 20% ανεργία, καταλαβαίνετε πόσο πολύ μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε, και η επιθυμία σας για προσωρινές κατηγορίες είναι και αυτό ενδιαφέρον για ενδιάμεσες. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι περιφέρειες, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη θα είναι κάθε ομάδα, δεν ξέρουμε τι μηχανισμούς θα έχουμε με το phasing in, phasing out Και έτσι δεν πρέπει να υποσχεθούμε υπερβολικά πράγματα τη στιγμή που ένα σωρό πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει. Να είμαστε δηλαδή σε μια μεταβατική περίοδο. Ούτε και οικονομικά πώς θα έχουν τα πράγματα. Τεχνικά λοιπόν, ωραία μεν που ξεκινάμε νωρί μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητάμε, αλλά απ' την άλλη προσοχή γιατί δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Έπειτα, για την στρατηγική της Λισαβόνας και για τη στρατηγική 2020. Η συζήτηση γίνεται στο Κοινοβούλιο και τον Ιούνιο στην Ολομέλεια θα υπάρξει ψήφισμα. Ελπίζω τουλάχιστον. Για τότε λοιπόν, όσον αφορά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, εγώ θυμάμαι τότε που είχαμε τον Κοκ που ήταν από τους πρώτους που αξιολόγησε αν μίλησε για τα προβλήματα, είπε ποιος πρέπει να ηγηθεί της όλης κατάστασης και τελικά έχει καταλήξει να είναι μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη ηγούνται του όλου εγχειρήματο. Και η αποτυχία της ε, Λισαβόνας είναι ακριβώς ότι οι αποκεντρωμένοι εταίροι, οι εταίροι οι οποίοι σε επίπεδο χωρών ή περιφερειών δεν έχουν συμμετάσχει αρκετά. Η Επιτρόπη των Περιφερειών είχαμε πει ότι έπρεπε να κάνει έλεγχο κάθε χρόνο να βλέπει ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά του στόχους και τα κριτήρια. Έγινε αυτό, αλλά επαναλαμβάνουμε τα ίδια σφάλματα. Και αυτό το λέω και στη συζήτηση, το είπα στην προηγούμενη Ολομέλεια όταν συζητήσαμε για τη στρατηγική 2020, πρέπει αποκεντρωμένα στην Ευρώπη να δούμε αυτά τα πράγματα. Είτε πρόκειται για μεγάλες πόλεις, είτε πρόκειται για νησιά, είτε πρόκειται για αγροτικές περιοχές, πρέπει όλοι αυτοί οι εταίροι να συμμετέχουν και να έχουν την ευκαιρία να πούνε την άποψή του. Η συζήτηση γίνεται στα κράτη-μέλη. Εγώ ξέρω τι γίνεται στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία ένα τεταρτάκι μιλήσαμε στην ε, Βουλή για τη Λισαβόνα και μετά είπαμε, ωραία, πάμε παρακάτω, πολύ ωραία, περνάμε στο επόμενο. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Όταν όμως αλλάζουν τα πράγματα και όταν έχουμε τα κείμενα της Επιτροπής, κοιτάξτε τα, πρόκειται για επικοινωνία εδώ. Μιλάει για επικοινωνία με τις αποκεντρωμένες ε, περιφέρειες. Μα είναι φοβερό να μην το κάνουμε, αφού το λέει. Η ιδέα σας λοιπόν είναι ακριβώς η αντιμετώπιση να είναι εδαφική. Όλες οι περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει να έχουν την ευκαιρία, να τους δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Εγώ ευχαρίστως συνυπογράφω και θέλω να τη δω αυτή τη δέσμευση από όλες τις πλευρές. Ώστε να βοηθήσουν όλοι να διαμορφωθεί η στρατηγική 2020. Αυτό το στηρίζω λοιπόν. Και το λέω και στις άλλες πολιτικές ομάδες. Στην επόμενη ολομέλεια θα έχουμε το ψήφισμα για τη στρατηγική 2020 και να συμπεριληφθεί και αυτό. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Σνάιντερ, σας ευχαριστώ θερμά για την ε, έκθεσή σας. Γνωρίζω εδώ και καιρό αυτή τη γνωμοδότηση και οφείλω να ομολογήσω ότι η συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή των Περιφερειών και που συνεχίζεται έχει αλληλεπίδραση με τη δική μας συζήτηση και διαπιστώνω ότι σε πολλά σημεία καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιφερειών. Συμφωνώ με τον κύριο Βανίστερ Ρόι ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η πολιτική συνοχής να μην γίνει ένας απλός προϋπολογισμός που θα εξυπηρετεί τη στρατηγική του 2020. Δεν είναι σαφές αυτό. Προς το παρόν τα διαρθρωτικά κονδύλια Μέχρι το 2013 εξυπηρετούν ε, την στρατηγική της Λισαβόνας. Μια στρατηγική που έχει αποτύχει και που δεν έχει διορθώσει τα προβλήματα. Και δεν μπήκαμε ακόμη στον κόπο να αναλύσουμε τις αδυναμίες της στρατηγικής της Λισαβόνας και πού πήγε στραβά και τι πήγε στραβά. Επίσης, και για την πολιτική της ε, συνοχής υπήρξαν κάποια προβλήματα. Και πριν κάνουμε την διεξοδική ανάλυση και την αξιολόγηση της προηγούμενης περίοδου μας προτείνουν μια νέα δεκαετή στρατηγική που θα ξεκινήσει το 2014. Βέβαια χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο. Και πριν ακόμη τη λήξη της περίοδου χρηματοδότησης πρέπει ήδη να λάβουμε απόφαση για την επόμενη περίοδο δεν είναι κακό να προετοιμαζόμαστε, αλλά δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Η πολιτική συνοχή είναι αυτόνομη πολιτική, ξεχωριστή. Καλό είναι να υπάρχουν συνέργειες με άλλες πολιτικές, αλλά δεν θα πρέπει να αντιστρέψουμε είναι να υποβαθμίσουμε τους στόχους της ε, πολιτικής συνοχής. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που δεν εξετάστηκε από την ε, Επιτροπή Περιφερειών και δεν περιλαμβάνεται στην γνωμοδότησή σας. Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες συζητούμε αυτό το θέμα του μέλλοντος της πολιτικής συνοχής και διαρωτόμαστε αν θα χρησιμοποιηθούν κυρώσεις από το Ταμείο Συνοχής απέναντι στα κράτη-μέλη που καταστρατηγούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους εφαρμόζουν ε, ατελώς. Ποια είναι η θέση της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής των Περιφερειών για το θέμα των κυρώσεων. Θα είναι σημαντική για τη διαμόρφωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έξι αγορητές είναι γεγραμμένοι στον κατάλογο. Τον ολοκληρώνω εδώ. Δεν θέλω καν να σας κοιτάξω για να αποφύγω προβλήματα. Αλλά μόνο 20 λεπτά μας έχουν απομείνει πριν την έναρξη των ψηφοφοριών, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αρκετά πειθαρχημένοι στη χρήση του χρόνου. Η Ελίζαμπετ Σρέτερ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν μια διευκρίνηση για την γνωμοδότηση. Σε μία σελίδα αναφέρεται μία θέση του ΕΛΚ. Είναι θέση του ΕΛΚ όμως ή της ε, Επιτροπής των Περιφερειών ολόκληρης. Γιατί συζητήσαμε τις θέσεις και τις απόψεις των ομάδων και η δική μας θέση απάδει της θέσης του ΕΛΚ. Και θα ήθελα να γίνει μια διευκρίνηση στο σημείο αυτό. Πώς να εκλάβουμε τον τίτλο ε, της γνωμοδότησης. Δεύτερον, κάτι που παραλήθηκε είναι ένα κέριο ζήτημα, το οικονομικό. Τα κονδύλια, ο προπολογισμό και η κατανομή των κονδυλίων γιατί είναι καλό να προσφέρουμε κάτι σε όλες τις περιφέρειες και ακούγεται και πολύ ωραία και αυτό προβλέπει η διαπεριφερειακή συνεργασία. Υπάρχουν κάποια πειραματικά προγράμματα και γνωρίζουμε το ύψος των κονδυλίων. Και δεν πρόκειται μόνο για προγράμματα της πολιτικής συνοχής, αλλά για πειραματικά προγράμματα, με πειραματικό επίσης και δοκιμαστικό προϋπολογισμό. Αλλά δεν αναφέρεται το θέμα της κατανομής αυτών των κονδυλίων. Ούτε έγινε καθόλου λόγος για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι το γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες έχουν το 60 ή το 75% ή μάλλον αυτές οι περιφέρειες κατά 60-75% δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν τους ε, στόχους. Και εξαιτήσεις της προσημείωσης της στρατηγικής της Λισαβόνας ε, είναι πολύ περιορισμένες στις δράσεις τους. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν επικριτική η Επιτροπή των Περιφερειών στο θέμα αυτό. Γιατί η πολιτική συνοχή είναι αυτόνομη πολιτική, έχει δική της αξία. Παρόλο που μερικές φορές ε, υπάγεται στη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρόκειται για κοινή απόφαση μεταξύ των ε, εθνικών κυβερνήσεων και των οργάνων της Ένωσης. Αλλά φαίνεται ότι οι αποφάσει λαμβάνονται από το πάνω προς τα κάτω. Είναι λοιπόν η Επιτροπή των Περιφερειών σε θέση να προβάλλει αυτές τις θέσεις, να αναπτύξει αυτή την πολιτική, να βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση από τη βάση προς τα άνω. Αυτό που ονομάζουμε bottom-up. Και αυτό που είχαμε ζητήσει και με την έκθεση ΒΑΚΑ. Ευχαριστώ. Uh, ε, ο τελευταίος ομιλητής τώρα και μετά έχουμε για τον πρώτο γύρο και μετά έχουμε άλλους τέσσερις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Σνάιντερ. Συγχαρητήρια για την γνωμοδότησή σας καταρχήν και για την παρουσίασή σας που ήταν πολύ αξιόλογη. Εγώ θα αναφερθώ στην παράγραφο 44 της γνωμοδότησής σας που προβλέπει το εξή. Θα πρέπει να, να θεσπιστούν τα κατάλληλα και δίκαια μεταβατικά προγράμματα ε, χάρη της σύγκλησης προκειμένου όταν έχει υπο... ξεπεραστεί το κατόφλι το 65% το 75% να δώσουμε ενισχύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες για να μην ε, μειωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Επίσης, θα πρέπει και στις περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στο 75% να δοθούν κάποια ειχέγγυα και μεγαλύτερη σταθερότητα για την ανάπτυξή τους. Εγώ προέρχομαι από μια υπεραπόμακρη περιοχή, την ίσο της Μαδέρας, που τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης από τη συνθήκη. Και εξαιτία ε, των αντίξεων καιρικών συνθήκων και της γεωγραφικής θέσης ε, χρήζει τέτοιας ε, ειδική και προνομιακή μεταχείριση. Γιατί θα πρέπει να προβλέψουμε ίση μεταχείριση για παρόμοιε πραγματικότητε και διαφορετική για καταστάσει που είναι πολύ διαφορετικέ. Όταν η Πορτογαλία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γύρω στο 45% του κοινοτικού μέσου όρου. Και μέσα στα 25 χρόνια πέρασε από το 40% του κοινοτικού μέσου όρου στο 95-96% του κοινοτικού μέσου όρου η Μαδέρα. Αυτό το διαπιστώσαμε όχι μόνο στη Μαδέρα αλλά και στα Κανάρια νησιά που είναι μια αυτόνομη περιοχή της Ισπανίας και που έχει υψηλό ΑΕΠ. Βρίσκεται και η περιοχή αυτή στο 98% του κοινοτικού μέσου όρου. Αλλά υπάρχουν προβλήματα άσχετα με την οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιφερειών. Γιατί η δυσκολία σε αυτών των ε, περιφερειών οφείλεται στη γεωγραφική τους θέση και στις ε, αντικσότητες που τους επιβάλλει η φύση. Οπότε δεν αρκεί οικονομική ε, αντιμετώπιση για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της φύσης. Και μάλιστα αυτή η περικοπή δραστική του προπολογισμού δημιουργεί προβλήματα και στα Κανάρια και στη Μαδέρα. Μεταξύ του 2000 και 2006 η Μαδέρα έλαβε από τον κοινοτικό προπολογισμό 1,98 δις. 1,098 δις και μάλιστα τελευταία περάσαμε από 1 δις 98 σε 730 εκατομμύρια ευρώ. Στις 20 Φεβρουαρίου, όπως ξέρετε, η Μαδέρα πλήγει από μια τρομακτική θεομηνία που προκάλεσε ζημίες ύψους ενός δις 70 εκατομμύριων. Μέσα σε έξι ε, ουσιαστικά ώρες καταιγίδα χάθηκαν όλα τα επιτεύγματα που υλοποιήθηκαν χάρη στα κοινοτικά κονδύλια μέσα σε μία εξαίτια. Είναι αναφυσβήτητο βέβαια ότι το ΑΕΠ είναι, αν όχι το μοναδικό, ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια που θα λάβουμε υπόψη για την κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων. Μήπως όμως θα πρέπει να εμπλουτίσουμε τον ΑΕΠ και με άλλους δείκτες. Στα Κανάρια, για παράδειγμα, σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο ποστό ανεργίας από όλε τι αυτόνομε περιοχέ τη Ισπανίας. Παρόλο που τα Κανάρια έχουν ΑΕΠ 98% του κοινοτικού μεσουόρου, έχουν 28,5% ε, ποσοστό ανεργία. Δηλαδή η κοινωνική κατάσταση στα Κανάρια βρίσκεται ουσιαστικά στο χείλο ε, της κοινωνική επανάσταση. Αλλά και στη Μαδέρα, την τελευταία τετραετία, η ανεργία διπλασιάστηκε, υπερδιπλασιάστηκε. Οπότε δεν αρκεί το ΑΕΠ. Θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλους δείκτες, όπως συμπεριλήψη νέων τεχνολογιών, το ποσοστό ανεργίας. Να συνοδεύσουμε το ΑΕΠ με άλλους δείκτες, να μην το θεωρήσουμε ως το μοναδικό δείκτη για την κατανομή των διαφορετικών κονδυλίων. Δεν αρκεί το ΑΕΠ. Ευχαριστώ και το λόγο κύριε Σνάιντερ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρο και ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι θα προσπαθήσουμε φυσικά να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, όταν με ρωτήσατε τι είναι η γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση επιτρέπει των περιφερειών είναι. Διαφορετικός, διαφορετικά δεν με είχατε καλέσει. Αυτό που σας παρουσιάζω εδώ, αυτό μάλλον που σας διανεμήθηκε εδώ δεν ήξερα ότι έχει διανεμηθεί. Πρόκειται για ένα έντυπο ε, το οποίο φαίνεται ότι ε, δημοσίευσε η πολιτική μου ομάδα με την έκθεση αυτή. Είναι μια πολιτική επιλογή, αλλά δεν είναι αυτό οι παρουσίες που σας κάνουν εδώ είναι της πολιτικής της Επιτροπής των Περιφερειών. Φυσικά το κείμενο της, της, της πολιτικής μου ομάδας πολύ ευχαρίστω να το δώσετε και παραπέρα. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συγκεκριμένα. Ε, προφανώς και στηρίζουμε τις θέσεις που περιλαμβάνονται μέσα στο έντυπό μας και στην γνωμοδότηση. Ω πρόεδρο τη ομάδα ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο στην Επιτροπή των Περιφερειών, πάντω με χαρά μπορώ να σα πω ότι οι συμβασμοί στου οποίου καταλήξαμε μέσα στην έκθεση αυτή είναι τόσο καλοί και τόσο συνεπεί που στέκουν ως συμβιβασμοί, στέκουν μέσα στη γνωμοδότησή μα. Προπολογισμό τώρα και διαθέσιμα κονδύλια. Είχαμε πει εξ αρχής ότι έχουμε βάσιμους λόγους να μην ε, διατυπώνουμε πιο συγκεκριμένες απαιτήσει ως προς την πρικοδότηση, ως προς τον προϋπολογισμό. Ε, και μεγάλο τμήμα βέβαια των ευρωπαϊκών κονδυλίων θέλουμε να συνεχίσουν να διατίθενται στην ε, πολιτική της νοχής αυτό το λέμε ξεκάθαρα, αλλά πρέπει πάντοτε αυτό να γίνεται σε συνάρτηση του τι θέλουμε και τι μπορεί να προσφέρει Δεν δεσμεύουμε λοιπόν κανέναν, δεν δίνουμε συγκεκριμένα ποσά στις διεκδικήσεις μας ως προς τα κονδύλια. Τώρα, εάν πρέπει να κάνουμε όπως λέμε και, και το ένα πράτην και το άλλο μία φιένε, δηλαδή να προσπαθούμε και το bottom-up αλλά και το top-down ως προσέγγιση χρειάζεται να υπάρχουν το earmarking, είναι επί παραδείγματι ο προσδορισμός οροσίμων μέσα από την στρατηγική της Λισαβόνας για μας ε, στη δική μου περιφέρεια συγκεκριμένα δεν ήταν χρήσιμο. Ε, δεν το θα θέλαμε ως ε, στόχο της στρατηγικής συνοχής. Θα πρέπει δηλαδή όταν θέλουμε να αναπτυχθεί μια περιφέρεια να πανεβαίνουμε μόνο εκεί όπου προβλέπει η στρατηγική Λισαβόνα να ε, γίνεται η παρέμβαση. Από την άλλη όμως διαπιστώνουμε ότι ενισχύεται το earmarking, όλο και περισσότερα δηλαδή ορόσημα προσδιορίζεται και τελικά χάνουμε το όραμα της ε, πολιτικής συνοχής και των συγκεκριμένων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που μπορεί να προσφέρει η πολιτική της συνοχής. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε μια, όπως λέω, αρμονική προσέγγιση στην ε, προσπάθεια αυτή. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής, ότι στο έγγραφό μας ξεκάθαρα λέμε ότι πρόκειται για ένα θέμα του κομματιού τη σύγκληση, δηλαδή στην Επιτροπή των Περιφερειών και δεν υπήρξαν αντίθετε τροπολογίε επισημένω στην γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να μιλάμε για περιφέρειες οι οποίε ανήκουν στο, στους στόχους αυτή τη στιγμή τη σύγκληση και οι οποίε σε μεγάλο βαθμό οφείλουν την ανάπτυξή τους στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στην προσεχή περίοδο ξεπερνούν το όριο του 75% προς τα άνω. Γι' αυτό θέλουμε να παραμείνουν μέσα στους στόχους της συνοχής, να παραμείνει η στήριξή τους. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περιοχές που βρίσκονται άνω του 75%, 75 με 90% φερρυπίν, θα ενσωματωθούν σε ένα νέο στόχο στήριξης. Αυτό όχι γιατί θέλουμε συνέχεια να δούμε χρήματα, αλλά γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε τις επενδύσεις μας και να καταστήσουμε την ανάπτυξη αυτών των περιφέρειων αηφόρα. Οι δείκτες. Κύριε Τισέιρα, πρέπει να σας πω ότι ανεξαρτήτως της αρχιτεκτονικής που επιλέγετε, στόχος 1, 2, 3 κτλ. Έχουν τις ιδιωτερότητέ τους οι περιφέρειες. Υπάρχουν οι άκρους απομακρυσμένες, υπάρχουν οι νησιωτικές περιφέρειες. Και χωρίς να είναι το Σιλ της Γερμανίας ή η Μαγιόρκα της Πορτογαλίας, προβληματικές περιοχές έχουν ε, προβλήματα, δυσκολίες ιδιαίτερες λόγω ακριβώς της γεωγραφικής τους θέσεως ή γεωφυσικής τους καταστάσεως, ότι είναι νησιωτικές περιοχές κτλ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια ιδιαίτερη μνήμα και ιδιαίτερη στήριξη. Η Μαδέιρα έχει καταπληκτική πρόοδο να επιδείξει ο συνάδελφος από την ομάδα, ο πρόεδρος Σαρντίμ, έχει ήδη ε, επιδείξει και αποδείξει μάλλον αυτή τη σημαντική πρόοδο της ε, Μαδέρα. Ύστερα λοιπόν από πολλές συζητήσεις συμφωνούμε νομίζω και καταλήγουμε ότι δεν πρέπει να να αποκλείσουμε στόχους που είναι οικουμενικοί, οι οποίοι μπορούν να είναι κατανοητοί σε κάθε περιφέρεια. Και ω στόχο θα πρέπει βέβαια να έχουμε το ΑΕΠ για το χαρακτηρισμό της περιφέρειας, αν είναι δηλαδή ισχυρή ή μη. Ο κύριος στόχος, το κύριο συνομικριτήριο κριτήριο για τον προσδορισμό της περιφέρειας θα είναι το ΑΕΠ. Διαρθρωτικά ταμεία ως μέσον κύρωσης. Ήταν μια ερώτηση της κυρίας Κρέλ, νομίζω, αλλά μάλλον δεν με ακούει. Προσωπική μόνο απάντηση που να σας δώσω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν συστήσαμε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Θεωρώ ότι είναι αντιπαραγωγική η άσκηση τέτοιων κυρώσεων. Τα εθνωτικά ταμεία είναι μέσα τα οποία στόχο έχουν να στηρίξουν ε, διατηθέμενα μια περιοχή που έχει προβλήματα. Εάν δοθεί εντύπωση ότι είναι μόνο ανταμοιβή, που μπορεί κανείς να αφαιρέσει από κάποιον εάν ε, δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, τότε νομίζω ότι δεν έχουν επιτελέσει τα μέσα αυτά το έργο τους. Και άρα δεν μπορούν πλέον να διατεθούν με αυτή την έννοια. Προσωπική μου επαναλαμβάνω γνώμη, είμαι πεπισμένος ότι υπάρχουν άλλα μέσα κύρωσης, άλλος τρόπος να πιεστεί κανείς ώστε να επιτελεί το καθήκον του. Αλλά το να αποδυναμώσουμε τον αδύναμο ακριβώς εκεί που τον πονάει, ακριβώς εκεί που είναι αδύναμος, νομίζω ότι είναι αντιπαραγωγικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε παρά να παραβούμε λίγο το χρονοδιάγραμμά μας και να αρχίσουμε αργότερα την ψηφοφορία, γιατί δυστυχώς έχουμε ακόμη αρκετούς ομιλητές. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα προσπαθήσω λέει η κυρια Ντεμπρούν. Ορισμένα κράτη-μέλη που τίθεται έκαναν πολύ καλή χρήση των διαρθρωτικών ταμείων την περασμένη περίοδο ήταν η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Και ακούσαμε στη συζήτηση χθε με τον κύριο Άνερ και την Βερόνικα Γκάφε ότι οι ανισότητε παρόλα αυτά στι περιοχές αυτές μεταξύ των περιφερειών, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ε, επιτάθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Και το ίδιο ξέρω ότι συνέβη και στην Ιρλανδία. Χαίρομαι για τα συμπεράσματά σας που αναφέρουν τους στόχους ε, της πολιτικής συνοχής και την ε, εναρμονισμένη ανάπτυξη των περιφερειών και την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Πώς όμως θα το λάβετε υπόψη αυτό στη συζητήση σας για την επόμενη περίοδο. Αυτή την πληροφορία που λάβατε ότι χώρε που είχαν αξιοποιήσει τα διαρθρωτικά κονδύλια παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να μειώσουν ή να περιορίσουν τι ανισότητε μεταξύ των περιφερειών του. Πώ θα το λάβατε υπόψη για την επόμενη περίοδο, Γιατί η προσημείωση, ο προκαθορισμό των κονδυλίων για συγκεκριμένου στόχου είναι σημαντικό. Τι άλλο είδου συζητήσει θα έχετε για να λάβετε υπόψη και αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ. Κύριο Άλβες, θα ήθελα να συγχαρώ τον Μάικ Σνάιντερ και την Επιτροπή Περιφερειών για τη γνωμοδότησή του. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή, περιφέρεια του στόχου 1, της Αζόρες, με πολιτική, οικονομική και διοικητική αυτονομία. Και υπό αυτό το πρίσμα εξετάζω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να προσυπογράψω αυτό το έγγραφο και αν ήμουν στην Επιτροπή Περιφερειών θα το ψήφιζα κι εγώ. Αναφέρεται η ανάγκη αποφυγής της επανεθνικοποίησης, εγώ θα έλεγα αποφυγής και της επαναπεριφερειοποίησης. Ε, μάλλον επαναπεριφερειοποίηση, δηλαδή όχι αφαίρεση των εξουσιών των περιφερειών και συγκέντρωση στις α, ε, κεντρικές αρχές της ε, διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων και των κονδυλίων θα πρέπει ε, να πηγαίνουν ε, απευθείας στις περιφέρειες οι ενισχύσεις αυτές, γιατί είναι σημαντικές οι πολιτικές της σύγκλησης, αλλά το πιο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι πολιτικές προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να αξιοποιηθεί το δυναμικό αυτών των περιφερειών εν ώψη της στρατηγικής του 2020. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της εφιούς ανάπτυξης, ε, της αηφόρου και της συμμετοχικής ανάπτυξης στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συντονισμό των πολιτικών, όχι να υπαγάγουμε την πολιτική σύγκληση στη στρατηγική, αλλά να συνδυάσουμε όλες αυτές τις στρατηγικές και να ευθυγραμμίσουμε τους στόχους των περιφερειών με τους στόχους της πολιτικής συνοχής γιατί δυστυχώς οι πόροι σπανίζουν αυτή την εποχή. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται πιο ορθολογική και αποτελεσματική τους χρήση και αξιοποίηση. Ο κύριος ε, Μάρκους Πίπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Σνάιντερ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά τους μηχανισμούς κυρώσεων που θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχή, ενδεχομένω τα γεωργικά ταμεία. Είναι κάτι που συστήσαμε και χθε με τον κύριο Άνερ τη Επιτροπή. Δεν φαντάζομαι να μπορεί ένα κράτος επανειλημμένα να προσβάλλει τα κριτήρια της σταθερότητας, του Συμφώνου Σταθερότητας, εφόσον υπάρχουν βέβαια σαφείς και αποτελεσματικοί μηχανισμοί έλεγχη. Ένα ερώτημα για, την, για τον στόχο της μετάβασης που αναφέρατε νωρίτερα. Είπατε ότι υπάρχουν, κράτη τα οποία, ε, υπάρχουν περιφέρειες μάλλον, οι οποίες βγαίνοντας από τον στόχο αποκλείονται και θέλουμε να τις ε, καλύψουμε κάπως η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση ως στόχοι νομίζω ότι έχουν προχωρήσει ιδιαίτερο. Σε ορισμένες περιφέρειες μάλιστα βλέπουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία με την ανάπτυξη μεγάλων δικτύων μέσα από τα προγράμματα αυτά, ε, ε, δικτύων διαπεριφερειακών μέσα στην Ευρώπη. Και ίσως λοιπόν ορισμένες περιοχές που ακόμη μπορεί στη Δυτική Ευρώπη να θεωρηθούν σχετικά φτωχές έχουν χάρη στη δικτύωση αυτή, δει ενίσχυση των κονδυλίων που μπορούν να διεκδικήσουν. Σε αυτό τι έχετε να πείτε. Ευχαριστώ, Σον Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια στον κύριο Σνάιντερ για την εξαιρετική εκθεσή του. Πολύ σύντομα. Ο κύριος Φαν Ρόι είπε, νομίζω κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στην υπόθεση αυτή. Αυτές. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό και θετικό, διότι οι τοπικές αρχές είναι αυτές που γνωρίζουν καλύτερα τι συμβαίνει με περιοχές, εμπλέκονται δηλαδή επιτόπου με την ε, λήψη των αποφάσεων. Αλλά όχι μόνο αυτό, η μόνο δύο, είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τοπικές αρχές είναι πολύ μακριά από τη λήψη αποφάσεων. Λαμβάνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τοπικές αρχές δεν έχουν καμία εμπλοκή. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να έχουμε καλύτερη, περισσότερη επικοινωνία και συμμετοχή σε αυτές τις προτάσεις των τοπικών αρχών. Και νομίζω θα ήταν καλό να ενσωματωθεί αυτό στις προτάσεις. Δεύτερον, Συμφωνώ με άλλες παρατηρήσεις που ακούστηκαν ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε την ταξινόμηση και την αξιολόγηση των ε, περιφερειών. Το 75% επί του, ΑΕΠ, του μέσου όρου ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώ είναι καλή λύση και αποτελεσματική, αλλά δεν μπορεί να αρκεί μόνο αυτό. Ασφαλώ υπάρχουν και άλλοι παράγοντε. Νομίζω ότι αυτό υπενήχθη ο κύριο Σνάιντερ, που έχουν να κάνουν και με την απασχόληση ή αντίστοιχα την υποαπασχόληση και την ανταγωνιστικότητα που μπορούν να επιτρέψουν την καταγραφή της ισχύω μιας φέρειας και αυτούς θα πρέπει να τους συμπεριλάβουμε. Αν έχουμε παραδείγματι μια περιοχή η οποία έχει 20% ανεργίας, ανεργία. Ε, ε, ίσως είναι ότι έχει το επί του ΑΕΠ πάνω από το 75% αλλά μόνο περιορισμένη ε, αλλά έχει υψηλή ανεργία 10-15% τότε ασφαλώς θα πρέπει να την ε, λάβουμε υπόψη στους στόχους της συνοχής και να τη στηρίξουμε. Και στη δική μου την πατρίδα υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια αναθεώρηση του τι, του τι συζητούμε και τι ταξινομούμε ως περιφέρεια. Η στρατηγική της Λισαβόνας πιστεύω ότι είχε καλούς στόχους και δεν ε, μ' αρέσει να ακούω κάθε φορά που λένε όλοι «Α, ήταν λάθος στρατηγική της Λισαβόνας, απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας», χωρίς ποτέ να εξηγείται το γιατί απέτυχε, γιατί υπάρχουν και πολύ σημαντικές επιτυχίες που έχει καταγράψει η στρατηγική της Λισαβόνας. Ας γίνει λοιπόν μια ανάλυση, ας γίνει μια αντικειμενική και ουδέτερη ανάλυση, γιατί πολλά ήταν τα θετικά στοιχεία της στρατηγικής της Λισαβόνας και αυτά δεν έχουν υπογραμμιστεί επαρκώς. Εάν λοιπόν λέει κανείς ότι απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας, είναι σαν να λέει ότι έχουμε αποτύχει όλοι, ότι απέτυχε ο ίδιο εκείνο ο οποίο εκλήθη να εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική, να υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή στα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κανεί σε τελευταία ανάλυση άμυρο ευθυνών. Δεν μπορούμε να λέμε ότι, για όλα, ότι όλα έχουν αποτύχει, ότι η στρατηγική τη Λισαβόνα ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Πρέπει να γνωρισουμε και τι επιτυχίε τη. Κύριε Στομόπουλο. Ήδη υπόθηκε ότι οι περιφερειακές ανισότητες σε κάποιες περιοχές ε, όπως την Ελλάδα αυξήθηκαν. Το χάσμα με τα νησιά, τις αστικές περιοχές και τις ε, μητροπολιτικές είναι πολύ μεγάλο. Με τι τρόπους μπορεί η πολιτική συνοχής να προσφέρει νέες επεξεργασίες και προσεγγίσεις στον περιορισμό αυτών των μεγάλων περιφερειακών ανισοτήτων και επίσης επειδή ένας από τους στόχους της, ε, της πολιτικής συνοχής στο μέλλον είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών και η ενίσχυση της επικουρικότητας. Με τι τρόπους θα μπορούμε να κρατούμε να κρατήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην επικουρικότητα και την παρακολούθηση της κατάστασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ja, Ο ähm, κύριος Σνάντερ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σημειώσω το εξής για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μιλούμε για προσδορισμό των περιφερειών με μόνο δείκτη ΑΕΠ και όχι άλλους δείκτες. Άλλοι δείκτες μπορεί να συζητηθούν αλλά σε άλλο επίπεδο, στην αξιολόγηση Φερρυπίν στο ζήτημα της, αξιολογιο... της ευελιξίας που μπορεί να έχει μια περιφέρεια. Αλλά για τον προσδιορισμό των περιφερειών φρονούμε εμείς ότι θα πρέπει να είναι μόνο το ΑΕΠ ο δείκτης που θα χρησιμοποιηθεί. Δεύτερον, μέσα για το στόχο 2. Κύριε Πίπερς, Ας προσπαθήσω να διατυπώσω τις θέσεις μου κατά τρόπο διπλωματικό. Εσκεμένα αποφύγαμε στην γνωμοδότηση την συγκεκριμένη αναφορά στην πρικοδότηση των στόχων, γενικά της πολιτικής συνοχής, πολλό δε μάλλον των συγκεκριμένων στόχων. Γι' αυτό και θα αποφύγω να κάνω οποιαδήποτε τέτοιου τοποθέτηση. Πάντως, δεν ήθελα να πω ότι θα πρέπει αποκλειστικά να πρόκειται για τι περιφερειέ τη τωρινή σύγκληση. Αυτόν τα προβλήματα δηλαδή περιγράφονται εδώ και αντίστοιχα με τον προπολογισμό και με τα δεδομένα τη σύγκληση που έχουμε αυτή τη στιγμή, χωρί να μιλούμε για ενίσχυση για, τη, για, τους, για τον τομέα αυτών προχωρούμε στην, στον προσδοσμό τη χρηματοδότηση. Για το ζήτημα των κυρώσεων ή την ε, έξοδο από το ταμείο, τα διαφορετικά ταμεία ε, ως, ως κύρωση, πρέπει να πω ότι υπάρχουν βέβαια διαφορετικές θέσεις στην υπόθεση αυτή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το να λέμε ε, υπήρξαν καταχρήσεις στην ε, χρήση των κονδυλίων ε, και ως εκ τούτου κλείνουν οι κρουνοί, σταματάει η χρηματοδότηση από τα διαφορετικά ταμεία, ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε μόνο γενικά ή μη τι άλλο, πάντως όχι ειδικά για τα διαφορετικά ταμεία. Ίσως θα είναι αυτό ένας ε, παράγοντας, μια λύση που θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε γενικά για κονδύλια του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, Φερρυπίν. Η στρατηγική Ευρώπη 2020, στρατηγική της Λισαβόνας τέθη ένα ζήτημα, να κάνω μια παραπομπή στα όσα είπε ο συνάδελφο Όλμπρεχτ πριν από μερικά χρόνια, σε σχέση με ακριβώ τη συνάφεια αυτή μεταξύ των δύο. Είχε πει λοιπόν ότι στη στρατηγική τη Λισαβόνα, που ήταν εκείνη την εποχή τη επικαιρότητα, είναι μια προσωρινή στρατηγική. Και αν όλα πάνε καλά, θα επιτευχθούν οι στόχοι τη Λισαβόνα, Οπότε θα πάψει να υπάρχει. Ξέρουμε το μεταξύ μα που δεν επιτεύξαν αυτή Και υπάρχει και η πολιτική τη συνοχή, η οποία είναι γεγραμμένη στην συνθήκη, αποτελεί δηλαδή βασική, μόνιμη και όχι προσωρινή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και για την εξέλιξη των κονδυλίων μέσα από τη στρατηγική του 2020. Είναι μια ad hoc στρατηγική η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο ω τέτοια μπορεί να ληφθεί υπόψη. Δεν έχει μονιμότητα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και βέβαια για τις, πολύ, για τις πολύτιμες παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά εκ μέρους όλης της Επιτροπής και προσβλέπουμε σε συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων. Και κάθε φορά που έχετε την αίσθηση ότι καταλήξετε σε πολύ σημαντική άποψη για το τι, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, καλό θα είναι να μας το κοινοποιείτε. Μας ενδιαφέρει πολύ τουλάχιστον. Περνάμε στις ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι, το σημείο 11 τη ημερήσια διάταξη, αλλά πρώτα να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να εξακριβώσουμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Βάλτε παρακαλώ τι κάρτε σας για να ελέγξουμε αν όλα τα μηχανήματα λειτουργούν. Vote is open. ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Again. Παρακαλώ μην μιλάτε. Συγκεντρωθείτε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Sorry, we are checking the machines. There is still people need to be Almost done. There is still somebody who who didn't vote. Yeah. I mean, not everybody checked. I think. Yeah can we close the vote? We close the Τέλος ψηφοφορίας. it works, no? Yeah, it works. It looks like it works. So we start with... Μάλλον λειτουργεί το σύστημα, οπότε περνάμε στην ψηφοφορία του σημείου 11, την έκθεση Σον Κέλλη. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Η Κωνσταντσα Κρέλ ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα παρακαλώ να υπολογιστεί η ψήφος του κυρίου Ολέντσεκ γιατί δεν έχει τη θέση του, δεν έχει συγγνώμη την κάρτα του, είναι όμως τη θέση του καθισμένος, ε, ψηφίζει τη δική του έκθεση, τουλάχιστον δείξτε κατανόηση, ανθρώπινα τα λάθη. Yes, please eh? speak up. I'm sorry, but I'm in the same position. Και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Έχω ξέχασα την κάρτα ψηφοφορίας. Μπορείτε να υπολογίσετε την ψήφο μου. Θα σηκώνω το χέρι, παρακαλώ. It's up to me, apparently. Ο πρόεδρος αποφασίζει, δεν έχω αντίρρηση. Θα συνυπολογίζουμε και τη δική σας ψήφο. Αλλά ελπίζω οι υπόλοιποι να έχουν φέρει τις κάρτες τους. Α, και κάτι άλλο, συνάδελφοι. Είναι πολύ δύσκολο για μας, γιατί δεν κάθεστε ανά Οπότε είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οπότε μην ξεχνάτε να σηκώνετε τα χέρια σας για να είναι σαφές το αποτέλεσμα. Γιατί οι περισσότερε ψηφοφορίε δεν θα γίνουν ηλεκτρονικά. Τροπολογία 1 Σον Κέλλη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται από ό,τι βλέπω. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 41 ψήφισαν υπέρ. Μία ψήφος, καμία αρνητική ψήφο και μία αποχή. Ωραία, συγχαρητήρια κύριε Σονκέλη και περνάμε στο σημείο 12. Το σημείο 12 είναι η έκθεση της κυρίας Ρόδη Κράτσα. Πολλές τροπολογίες συνάδελφοι, οπότε παρακαλώ να είστε συγκεντρωμένοι. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά τη γνώμη μου εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές κατά τη γνώμη μου έχει εγκριθεί τροπολογία 31 υπέρ καταπίπτει καταπίπτει 31 συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Αβέβαιο το αποτέλεσμα, ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται 20 ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν το δεύτερο τμήμα της 35. 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές κατά τη γνώμη μου έχει εγκριθεί. Την τροπολογία 52 δεν θα την ψηφίσουμε γιατί είναι γλωσσική. Πάμε στην 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίθηκε και η 53. Καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την, για την τροπολογία 53 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία, 31 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, τρέπεται εδώ το Πρόεδρο που το κατάλαβε, 54 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία η 59 καταπίπτει. 62. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 με προφορική τροπολογία όπως έχει τροποποιηθεί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Νέα αιτιολογική σκέψη με προφορική τροπολογία της κυρίας Κράτσα. Δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ποιο είναι υπέρ της τροπολογίας 1 για την αιτιολογική σκέψη α, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το σε, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη σε α, νέα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ολόκληρη την έκθεση ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος, ψήφισαν 42 υπέρ, κανένας κατά και δύο εποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Κράτσα. So we go now. Τώρα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε, τελειώνει εδώ αυτή η ψηφοφορία και περνάμε στο σημείο 13 που είναι η έκθεση του κυρίου Λινίτσεν για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Εδώ έχουμε πολλές τροπολογίες, θα είναι μακρά η ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν, είσαστε όλοι έτοιμοι. Ωραία, συμβιβαστική αριθμός 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Με προφορική τροποποίηση. Δεν έχετε αντίρρηση για την προφορική τροποποίηση. Ωραία, την τροποποιημένη τροπολογία λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόκειται για την τροπολογία αριθμός 11. Με τροποποίηση. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 24 κατά. Τώρα, συνάδελφοι, ψηφίζουμε την τροπολογία 11, χωρίς την τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπάρχει και εδώ προφορική τροποποίηση. Αντιρρήσεις για την προφορική τροποποίηση. Ναι. Ο κύριος Όνιτζακ. Α, οπότε δεν μπορούμε να διδεχτούμε την προφορική τροποποίηση. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Της ΕΝΒΙ τώρα, 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110. Τροπολογία 110. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε τροπολογία 5 της Επιτροπής Περιβάλλοντος Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 49. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. 1. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την τροπολογία 53 με προφορική τροποποίηση. Δεν έχετε αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση, όχι. Ωραία. Με την τροποποίηση λοιπόν ψηφίζουμε τροπολογία τρία. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Εγκρίνεται. 54 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε περνάμε τώρα στην τροπολογία 63. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατά τη γνώμη μου. Αν θέλετε να το ελέγξουμε. Ωραία. 65. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 65. Ξεκινάει η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 23 κατά. Απορρίπτεται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 Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. 27 υπέρ και 18 κατά. 78. Όχι. Διορθώνει η πρόεδρος. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα 79 με κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν ξέρω, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. 82 ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 82. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22-18. Τώρα, τροπολογία 84. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα 13 συμβαστική υπέρ, υπέρ της συμβαστικής 13, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία, α όχι, 14, συμβαστική 14 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται η συμβαστική 16. Τροπολογία 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 109 με προφορική υπέρ, κατά. Α, ο κύριος Σολενίτσιον έχει αντίρρηση. Είστε κατά Είστε κατά. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα στην προφορική τροπολογία να προσθέσουμε κάτι. Δηλαδή, δεσμεύει τον πρόεδρο να διαβιβάσει την, το ψήφισμα στο κοινοβούλιο, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ρωσική Ομοσπονδία, τη Λευκορωσία και την Ορβηγία. Θα ήθελα έτσι να συμπληρωθεί η προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην τροποποίηση αυτή, στην τροπολογία 109. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε λοιπόν την διπλά τροποποιημένη τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία, οπότε έχουμε αυτή τη διπλή τροποποίηση, εγκρίθηκε. Τώρα τα αιτιολογικά. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά δεν ξέρω. Να ελέγξουμε καλύτερα. Ετυλογική σκέψη Β, τροπολογία 3. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίθηκε. 26 υπέρ, 20 κατά. Δέλτα, τροπολογία 6. Έχουμε μια προφορική τροποποίηση εδώ. Ψηφίζουμε, έτσι. Ετυλογική σκέψη δέλτα, τροποποιημένη, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Νομίζω και εσείς το νομίζετε, οπότε εντάξει. Ευχαριστημένο το ΕΛΚ, λέει η Πρόεδρος. Κερδίσατε, αλλά θέλετε να ψηφίσουμε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Τροπολογία 6 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία με την τροποποίηση της τροπολογίας 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 29-15. Είστε κατά. 29-16 τότε. Εγκρίνεται όμως παρόλα αυτά. Τώρα, ΑΦΕΤ 2. Εδώ έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα. Αφέτ 3. Πάλι κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αφέτ 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αφέτ 7. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Αφετ 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αφετ 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αφετ 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στις προτάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος. 1. Υπέρ, κατά, αποχές Ένβι NV2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. NV3 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε. Ωραία, θα ελέγξουμε για την τροπολογία 3 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. 23-21 εγκρίνεται. NV4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NV6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. NV7 υπέρ, κατά, Αποχές δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά με τους σοσιαλιστές, δεν ξέρω τι. Πρέπει να ελέγξουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την τροπολογία 7 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 21 κατά. Αυτοί που δεν ψήφισαν δεν θέλουν να ψηφίσουν τώρα τίποτα, να προσθέσουμε την ψήφα τους. Όχι. Καλά. Εγκρίνεται λοιπόν. Ένβη 11. Συνάδελφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Αν δεν θέλει το έλεγχο να ελέγξουμε. Α, να ελέγξουμε. Ωραία, 13. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, κατά τη γνώμη μου. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοιτάξτε, ας ελέγξουμε τη 16 για να είμαστε σίγουροι. Ηλεκτρονικός έλεγχος 16, ένβη. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορία. 23 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Και εδώ έχουμε την πρόταση αριθμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά τη γνώμη μου. 2 τραν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την πρόταση Επιτροπής Μεταφορών αριθμός 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας προφορίας, 21 ψήφοι υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 7. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τραν 7. Ψηφίστε. Πέρας της προφορίας. 23 υπέρ, 22 κατά. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα από εδώ. 8 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε Ηλεκτρονικό έλεγχο για την πρόταση επιτροπή Μεταφορών αριθμό 10. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορία, 25 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Ακόμα και αν ψηφίσουμε την ψήφο σα. 11 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές δεν ξέρω. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρόταση 14 της Επιτροπής Μεταφορών. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες 25 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Θέλετε να ελέγξουμε. Ή ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15. Ψηφίστε παρακαλώ. 22 υπέρ, 21 κατά. 16 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 17. Ψηφίστε παρακαλώ. 17 τραν. ...26 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο της ε, έκθεσης, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Ολενίτσακ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Λάσλο είναι εδώ. Μάλιστα, περνάμε στο σημείο 14. Θέλω να δώσω το λόγο στον εισηγητή Λάσλο Σούριαν για να μας εξηγήσει τις διαδικασίες του προπολογισμού. Είναι το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι, και το λόγο έχει Λάσλο Σουριάν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φαίνεται ότι είναι πολλοί συνάδελφοι που φεύγουν, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ενδιαφέρον ο προπολογισμό σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ουγγρικά. Περιμένω να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας. Kedves kollégák, az első feladatom talán az, hogy elmondjam πρώτο αρχικό μου καθήκον είναι να σας πω ποιες είναι οι συνθήκες με τι οποίες ξεκινά αυτή η διαδικασία για τον προϋπολογισμό. Έχουμε τώρα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ε, την οποία θέλουμε να πραγματοποιήσουμε σήμερα. και νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε ε, την πρακτική που είχαμε και σε προηγούμενα έτη. Λίγο πολύ το ίδιο δηλαδή σύστημα και βέβαια άκρος σημαντικό είναι τώρα ε, να είμαστε προετοιμασμένοι εγκαίρως, να έχουμε εγκαίρως το κείμενό μας έτοιμο και φυσικά η, τωρινή, η σημερινή ανταλλαγή απόψε αποτελεί την προετοιμασία του αρχικού κειμένου. Στη συνέχεια θα περάσει αυτό στη μετάφραση μέχρι τις 12 Ιουλίου, δηλαδή μέσα σε πέντε εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία έτσι ώστε η Επιτροπή να δει το κείμενο ε, στην ε, πλήρη του μορφή. Τώρα, όπως είπα, μόνο ανταλλαγή απόψεων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Τον Ιούλιο θα έχουμε το πλήρες κείμενο, το τελικό κείμενο. Και τέλη Ιουλίου, από ό,τι μας λέει η Γραμματεία μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε δύο εβδομάδες συγκεκριμένα μετά την υποβολή της τελικής μορφής της εκθέσεως στην Επιτροπή, να ορίσουμε την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Προθεσμία την οποία θέλω εξάπαντος να τηρήσουμε, διότι χρειαζόμαστε τέσσερες ημέρες για την λήψη αποφάσεως σχετικής με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Απόφαση η οποία θα ε, αλλάξει ουσιοδός τα, ε, την κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται η δημοσιονομική μας διαδικασία. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, υποβάλλεται αυτή η πρόταση. Και ασφαλώς θα χρειαστεί στην πρόταση αυτή να κατευθούν τροπολογίες, δεν υπάρχει εμφολία σε αυτό. Βέβαια πρέπει να επισημάνω ότι αυτό δεν είναι δικό μου τόσο καθήκον, όσο μάλλον μια, ένας αυτοματισμός, αν θέλετε, της ε, ε διαδικασίας, η οποία, ο οποίος προσπαθεί να ανατρέψει περικοπές που έχουν γίνει στην πρόταση. Άρα λοιπόν έχουμε προς το παρόν, όπως είπα, μόνο το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έχουμε το κείμενο της Επιτροπής, το κείμενο του Συμβουλίου, τα δύο, τα δύο έγγραφα αναφοράς, πάνω στα οποία στηριχθήκαμε και στις 6 Νοεμβρίου, Ιουλίου, συγγνώμη, θα κάνουμε τις, ε, τρο, στο Το Σεπτέμβριο μάλλον θα γίνει η τελική τροποποίηση του κειμένου. Έχουμε χρόνο δηλαδή αρκετό μέχρι το φθινόπωρο. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει την ψηφοφορία της εγκαίρως, πριν από την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου δηλαδή, άρα υπάρχει επαρκή χρόνο για συζήτηση, για ψηφοφορία και βεβαίω καλό θα είναι το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ψηφίσει στις 18 Σεπτεμβρίου έτσι ώστε μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου να γίνουν οι πρώτες φάσεις, να λάβουν χώρα οι πρώτες φάσεις της διαβούλευσης, όπως ορίζει η νέα διαδικασία. Τώρα, μου επιτρέπετε, να κάνω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχετικές με τον κανονισμό και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Η εικόνα που μας δίνει η πρόταση της Επιτροπής. Έχουμε γενικά μια καλή εικόνα στο τμήμα 1β έχουμε μία ε, αύξηση των κονδυλίων κατά 17%. 2007, 2008, 2009 ήταν έτη κατά τα οποία η πολιτική της συνοχής, ιδιαίτερα τα κονδύλια της ε, πολιτικής συνοχής ως προς τις δαπάνες, παρουσίαζαν μία στασιμότητα, κυρίως σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, και έτσι στο δεύτερο ήμιση του κύκλου, γιατί έχουμε φτάσει πια να συζητούμε τον προπολογισμό του 2011 και μετά βεβαίως το 2012-2013 έπονται, ε, όπου περιμένουμε ενίσχυση ως προς τις δαπάνες των προβλέψεων. Και άρα αυτό το 17% που προβλέπεται ως αύξηση των κονδυλίων ίσως να μην ε, αποδεχθεί επαρκές. Η συζήτηση που γίνεται κάθε χρόνο με το Συμβούλιο ασφαλώς θα επαναληφθεί και φέτος και θα δούμε τι θα προκύψει από αυτήν. Φυσικά ελπίζω ότι θα έχω την υποστήριξη της Επιτροπής μας για την ε, τοποθέτησή μου ως προς το ότι θεωρούμε ότι δεν επαρκεί για και δεν αντιστοιχεί στις ε, δαπάνες αυτή η αύξηση. Τώρα αυτό ήταν η θετική προοπτική, αλλά έχω και κάποια αρνητικά πράγματα να σας αναφέρω σε σχέση με το τμήμα 1β, συνοχή, ανάπτυξη, απασχόληση. Έχουμε αύξηση της τάξης του 3,6%. Σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι στο Ταμείο Συνοχής έχουμε αυξημένες ανάγκες και όχι αντίστοιχη αύξηση της πρικοδότησης. Και ως εκ τούτου προκύπτει ξεκάθαρα πως τα κράτη τα οποία αφορά ε, το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κονδύλια ενώ εφέτος, στην αρχή του χρόνου, το Μάρτιο, ήταν η κατάσταση αρκετά δύσκολη και στις πιστώσεις πληρωμών βλέπαμε μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε λίγο πολύ ε, φτάσει στα μισά του δρόμου και δεν είναι κατά την άποψή μου σωστό ότι το Συμβούλιο έχει μια αρνητική τάση στην υπόθεση αυτή, μειώνει δηλαδή τα κονδύλια. Κατά τα άλλα όμως πιστεύω ότι θα πρέπει και η Επιτροπή των προϋπολογισμών μας να στρατευτεί, να αγωνιστεί για να διαφυλάξει την πολιτική, την περιφερειακή, την πολιτική της συνοχής και νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε κόκκινες γραμμές και να πούμε ότι αυτό και αυτό από τις προτάσεις του Συμβουλίου θεωρούμε ότι αποκλείεται να τα δεχθούμε. Δηλαδή να ορίσουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και να ε, ελπίσουμε ότι έτσι θα έχουμε μια καλύτερη στρατηγική. Γιατί η αλλαγή στρατηγικής πιστεύω ότι είναι απαραίτητη στη διαδικασία του προπολογισμού. Θα πρέπει να ε, συμπεριφερθούμε κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι, μέχρι τα, από τα τελευταία χρόνια, από ό,τι μέχρι τώρα. Αλλαγή στρατηγικής μπορεί να μα φέρει περισσότερες ελπίδε επιτυχία. Και θα ήθελα επίση να αναφέρω κάποιε ανησυχίε απευθυνόμενο φυσικά προς τις πολιτικές ομάδες ε, εκφράζοντας και τις δικές μου θέσεις και της πολιτικής μου ομάδας τις θέσεις, το εξής. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μερικές φορές έχουμε μετριοπαθείς διεκδικήσεις, ενώ έχουμε περιθώριο αρκετά μεγάλο. Φερρυπίν έχουμε συνολικά ποσά μεγάλα, ενώ το περιθώριο το οποίο ορίζουμε ε, είναι κάπου στα 60 εκατομμύρια, ίσως να μην είναι αρκετά σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ο κύριος και ο παλαιός συνάδελφος, ο οποίος ε, είχε και την ε, πρωτοβουλία από πλευρά τη στη διαδικασία αυτή πλέον, ε, μπορεί να, αποδειχθεί ε, χρήσιμος ε, σύμμαχος κάνοντας προτάσεις οι οποίες είναι πιο θετικές για αυτόν τον προϋπολογισμό. Για τα πιλωτικά προγράμματα όμως, βλέπουμε ότι θα βρεθούμε σε μεγάλη δυσκολία γιατί οι επαρκείς πόροι δεν προβλέπονται και θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε τις τροποποίησεις στις προσδοκίες μας. Και ίσως και να φτάσουμε σε σημείο ρήξη Συμβούλιο, Επιτροπή, Κοινοβούλιο, ως προς την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πέραν του Κοινοβουλίου κανείς δεν είναι διατηθειμένος να δεχτεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν ε, τα πράγματα και σε σχέση με την Επιτροπή των Περιφερειών. Όπως είπα, η χρονική αυτή διάσταση, τη χρονική συνιστόσα, μας φέρνει σε μία, στην υποχρέωση, στην προσοχή ολομέλη να λάβουμε απόφαση για το τι θα κάνουμε για τα ε, πολλά κονδύλια για δισεκατομμύρια ευρώ μιλάμε, τα οποία δεν διατέθηκαν από πέρυσι, αν θα μεταφερθούν και πώς θα μεταφερθούν και βέβαια να αποφύγουμε την τρογοπέδη που προσπαθεί να επιβάλλει το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε μέσα σε μεγάλη οικονομική κρίση, το καλύτερο μέσο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να την αντιμετωπίσει την κρίση είναι η πολιτική συνοχή. Γι' αυτό θα πρέπει να διαφυλαχθεί και γι' αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε τα κονδύλια να διατίθενται σωστά από τα κράτη-μέλη και να είναι κατάλληλα επαρκή τα κονδύλια που θα διατίθενται στο πλαίσιο αυτό της πολιτικής συνοχής. Φυσικά θα γίνουν δύσκολες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις σκληρές αναμένεται να αναπτυχθούν γιατί και τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία υποχρεούνται να περικόψουν σε σχέση με τον περσινό τους προπολογισμό τον φετινό τους ε, κατά 20%. Είναι λοιπόν δύσκολες οι περιστάσεις και δεν μπορεί κανείς να περιμένει να ε, αυξηθεί η πρικοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η Ισπανία, Φερρυπίνη, η οποία βρίσκεται σε δινή κατάσταση, κάνει περικοπές της τάξης του 50%. Ε, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη θα πρέπει παραδείγματι να λάβουμε υπόψη ότι τα, τα πλεονάσματα δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να, σε, να διατίθενται σε νέα σχέδια από την ε, εδαφική ανάπτυξη, από την περιφερειακή ε, ανάπτυξη, την συνοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια τα οποία χρειάζονται χρηματοδότηση από αυτά τα πλεονάσματα. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορώ να πω με αρκετή βεβαιότητα πως μας, μας ε, υποστηρίζει και ο Επίτροπος για τα πιλωτικά σχέδια. Για τα πιλωτικά σχέδια έχουμε συνεργαστεί αυτές τις τελευταίες ημέρες με τους συναδέλφους από τους οποίους ε, ζήτησα να με στηρίξουν, να συμμετάσχουν στην επεξεργασία της προτάσεως Και σημαντικό είναι εδώ η, ε, να, υπάρ, να, να τηρηθεί ε, η διοργανική συμφωνία, η συμφωνία που υφίσταται ήδη, η οποία μπορεί να μας καθοδηγήσει στον τρόπο αντιμετώπισης των πιλωτικών προγραμμάτων ή σχεδίων και να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι ακόμη για ποια προγράμματα ε, θέλει να ε, δώσει την προτεραιότητα, σε ποια προγράμματα θέλω να δώσω την προτεραιότητα, ποια θεωρεί άκρο απαραίτητο να προχωρήσουν σε υλοποίηση, ποια ενδεχομένω μπορεί να αποκλείσει ή προτιμά να αποκλείσει. Έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμεί να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εξετασία αυτή τη υπόθεση και μέχρι το, το φθινόπωρο να έχουμε έτοιμη τη γνωμοδότηση. Όπω είπαμε, υπάρχουν κάποια από τα πιλωτικά σχέδια τα οποία τα υποστηρίζει η Επιτροπή. Ενδεχομένω όμω θα πρέπει να γίνουν σχετικέ τροποποιήσει ή ε, διορθώσει στον προπολογισμό και η Επιτροπή θα προσπαθήσει βεβαίως ως Επιτροπή να παραμείνει στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Ε, δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή για πόσα εκατομμύρια ευρώ μπορούμε να μιλούμε. Καλό όμως θα ήταν να είμαστε εμείς έτοιμοι και να πούμε εμείς προκαταβολικά κοιτάξτε οι προτεραιότητες είναι αυτές. Εμείς θέλουμε εκεί να δώσουμε τόσα λεφτά. Ε, και ενδεχομένως από τον τάδε ή δύνατο τομέα να κόψουμε τη χρηματοδότηση. Δηλαδή να είμαστε εμεί έτοιμοι για να κάνουμε τι σχετικέ επιλογέ. Πρέπει να πω επίση ότι είμαι και μέλο τακτικό στην Επιτροπή των Προπολογισμών και μπορώ και από εκεί με την ε, ε, δουλειά μου και βέβαια με την επιμονή μου να πείσω να μας ακολουθήσουν στις δικές μας προτιμήσεις. Και αυτό το κάνω ούτως ή άλλως και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη δική μου γνωμοδότηση. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι για τα πιλωτικά σχέδια, όπως έχουν σχεδιαστεί ε, μέχρι τώρα, όπως έχουν χαραχθεί, αναμένεται να υπάρξει μια κάποια βελτίωση ε, μέσα από τη διαδικασία της ε, κατάρτισης και των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Βελτίωση πάνω απ' όλα όσον αφορά τον έλεγχο. Και δεύτερον, πρέπει να επισημάνω για τα πιλωτικά αυτά σχέδια ότι την σοβαρή, την τελική απόφαση την ε, λαμβάνουμε με την ψηφοφορία το φθινόπωρο. Αυτή είναι η ημερομηνία που όλοι πρέπει να σημειώσουμε και να μην την χάσουμε. Ιδιαίτερο σε αν έχουμε να συζητήσουμε σοβαρέ περικοπέ. Πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση. Και βεβαίω θα πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε τα χρήματα που θα ετεθούν να είναι επαρκή, να μην είναι ε, τόσο μικρή η πρικοδότηση που να μην έχει κανένα αποτέλεσμα και σε τελευταία ανάλυση μην ξεχνάμε ότι τα κονδύλια αυτά απορρέουν ε, από πολιτικές και προγράμματα εγγεγραμμένα στη συνθήκη. Επίσης πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα αυτά τα οποία από τον ε, Ευρωπαίο φορολογούμενο αντλούν και διαθέτουν στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό αξιοποιούνται σωστά. Πηγαίνουν και πιάνουν τόπο. Τα, τα κονδύλια του, του Ταμείου Συνοχής, των Διαγνωτικών Ταμείων είναι απαραίτητα για την ε, έξοδο από την κρίση. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να περικοπούν και γι' αυτό πιστεύω ότι εάν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση μπορούμε και θέσει εργασία να δημιουργήσουμε και να βρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την έξοδο από την κρίση. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα, όπως είπα, πραγματοποιούμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα περιοριστώ σε αυτές τις γενικές παρατηρήσεις από πλευρά. μου. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση και υπόσχομαι να λάβω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως από τους συναδέλφους. Φυσικά μπορούν ε, οι ομάδες ε, να ε, τοποθετηθούν μπορούμε να έχουμε και διμερείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε διαχωριστικές γραμμές των ομάδων. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή κάθε ομάδα να ορίσει τις δικές της θέσεις και να ε, μιλήσει μόνο με τέτοιους όρους. Νομίζω ότι είναι καλό πέραν των ε, πολιτικών ομάδων να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή θέση, ένα καλό έγγραφο. Είμαι πεπισμένος δε ότι δεν είναι μόνο η δική μου η πολιτική ομάδα ε, που έχει αυτή τη θέση, ούτε η δική μου εθνική αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν σε αυτό ότι χρειάζεται μια κοινή γνωμοδότηση ως προς τον προϋπολογισμό και σε αυτό νομίζω μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, μπορούμε να προσδιορίσουμε την ευελιξία αυτή ε, μέσα από το έγγραφο και να ε, δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε κύριε Λάσλο Σούριαν. Ζήτησαν το λόγο δύο συνάδελφοι. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μας έχει μείνει μόνο ένα τέταρτο ακόμη για το θέμα αυτό. Ο κύριος Γκοντουμάνης. Ζήτησα το λόγο γιατί είμαι μέλος και της Επιτροπής Προϋπολογισμών και χθε ψηφίσαμε μία πρόταση της κυρίας Χοφμάγερ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, μία τροπολογία που υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις χώρες που έχουν χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διαρθρωτικών κονδυλίων. Και μάλιστα το είπε και σε πολλούς συναδέλφους. Είναι εύκολο να βρούμε ποιες χώρες είναι αυτές που δεν απορροφούν επαρκώς τα διαρθρωτικά κονδύλια. Να πω όμως και δύο λόγια για τα χρήματα, για τον προϋπολογισμό. Πιο ειδικά σχόλια. Καταρχήν, η περιφερειακή πολιτική που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει θα λάβει 4 εκατομμύρια επιπλέον σε διοικητικές δαπάνες και η διοίκηση που ασχολείται με τα κονδύλια αυτά θα έχει λίγο παραπάνω από 4 εκατομμύρια. Για το 2009 είχαμε 87 εκατομμύρια. Φέτος 85 και του χρόνου θα έχουμε 89 εκατομμύρια. Κανένα δεν μπορεί να παραπονιέται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει αρκετά κονδύλια. Όλα τα ταμεία και το Περιφερειακό και το Ταμείο συνοχή. και δεν ξέρω τι ποσοστό είναι το 85, τα 85 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά το ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχουν μείνει κάποια κονδύλια από τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, του 2000-2006. Μειώνεται βέβαια το ποσό αυτό. Και ο στόχος 1 είναι από 2 δις 1,8. Αυτό μένει για να δοθεί από το ΦΕΝΤΕΡ. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο στόχος 2 δεν μειώνεται τόσο όσο ο στόχος 1. Για, όλες, για όλη την περίοδο έχουμε 437 εκατομμύρια για να καλύψουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές που έχουν περιοχές του στόχου 2 στο Περιφερειακό Ταμείο. Επίσης, θα πρέπει να διεκπαιρεωθούν και κάποια σχέδια, όπως το Urban, για τις πληρωμές και επίσης η Βόρεια Αρλανδία έχει ακόμη να λαμβάνει 50 εκατομμύρια. Οπότε, ο κύριος Σούριαν είπε ότι το περιθώριο είναι πολύ στενό δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί εμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι σωρεύσαμε τις πληρωμές και σωρεύσαμε και τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Αν δείτε όμως σε σωρευτική βάση, έχουμε στο αποθεματικό 110 δις. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να αυξήσει ε, τις πληρωμές, λαμβάνει το σωρευτικό αποτέλεσμα πληρωμές συν ανάληψη υποχρεώσεων και στις αρχές του 2007-2008 οι πληρωμές ήταν πολύ χαμηλότερες από τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Αλλά για το 2010-2011, για το Περιφερειακό Ταμείο, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είχαμε ανάληψη υποχρεώσεων 23,6 δις, ε, έναντι 22,7 δις για φέτος. Δηλαδή ένα περίπου δισεκατομμύριο περισσότερο και 4 δις περισσότερα για τις πληρωμές. 18 δις αντί για 14 δις. Αυτό είναι το τμήμα σύγκλησης του ΦΕΝΤΕΡ. Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και την απασχόληση, εκεί η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Εδώ οι πληρωμές είναι μόνο ένα δις περισσότερο από τη φέτος. Αν κάποιος αναλύσει τον προϋπολογισμό βλέπει ότι άλλο σχέδιο ισχύει για το στόχο 2 και άλλο για το στόχο 1. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά απορρόφησης, δεν είναι σαφές γιατί είναι μόνο 2% λιγότερο για το στόχο 2. Γιατί οι χώρες του στόχου 2 είναι πιο ανεπτυγμένες. Αλλά το ποσοστό απορρόφηση είναι χαμηλότερο στο στόχο 2 από ό,τι στο στόχο 1. Σε ό,τι αφορά τα πειραματικά προγράμματα, δίκαιο έχει ο κύριος Σούριαν ότι πολλά πειραματικά προγράμματα μπήκαν στο προσυπόμνηση για την περιφερειακή πολιτική. Ε, εντάξει το Ρωμά, έρασμος, διεύρυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας με την πρόθεση της περιφερειακής πολιτικής, προπαρασκευαστικές δράσεις για τη δημιουργία πρόσφορου κλίματος για τις μικροπιστώσεις και ούτω, καθεστη, ούτω καθεξής. Για να παραταθούν όμως αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία και να γίνουν κάποιες διατυπώσει, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής, η διαφορά μεταξύ ανάληψη υποχρεώσεων ε, για το 2010-2010 είναι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο, σε αντίθεση με το ΦΕΝΤΕΡ. Στο ε, Ταμείο Συνοχής έχουμε ένα 11 δις 073, ενώ φέτος είχαμε για το 2011, ενώ Πέρυσι είχαμε 10-180, 10 ε, και στις πληρωμές λίγο λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια. Θα δοθούν 6,2 στο 2011 αντί 4,3 φέτος. Φαίνεται ότι προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό στις πληρωμές που ήταν πολύ μικρό το ποσοστό του στην αρχή των δημοσιονομικών προοπτικών. Πάντως, εν γέννη, θα ήθελα να πω ότι θα γίνουν μάχες για τα κονδύλια αυτά και για το σύνολο της περιφερειακής πολιτικής, βλέπουμε ότι έχει 13 προγράμματα. Και εκεί βλέπουμε τις πληρωμές, οι περισσότερες πληρωμές για την περιφερειακή πολιτική για το 2011 θα είναι 18,1% σε σχέση με το 2010. Αν δείτε τις άλλες πολιτικές, δεν θα βρείτε τόσο μεγάλη αύξηση. Λίγες πολιτικές έχουν μεγαλύτερο ποσοστό. 27% για την ιστορική αγορά, αλλά εκεί είναι χαμηλότερα τα κονδύλια. Οπότε έχουμε 5 δις για τις πληρωμές. Δεν είναι δίκαιο να λέει κανείς ότι είναι ισχνά τα κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής, αλλά άλλες, περιφε... άλλες πολιτικές έλαβαν πολύ λιγότερα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Εκεί η αύξηση είναι μόνο 3,8%. Και αυτό το 3,8% όντως είναι μικρή αύξηση για την ανάληψη υποχρεώσεων. Επίσης θα ήθελα να σας δώσω ένα στοιχείο για να το θυμάστε. Αν δούμε όλες τις αλλαγές από το 2007 έως το 2017, πλην και τα συν, και για τις υποχρεώσεις και για τις ε, πληρωμές και τα αθροίσετε όλα αυτά, συγκρίνεται το 2007 και το 2011. Δύο στοιχεία θα σα δώσω για να το θυμάστε. Στις, στην ανάληψη υποχρεώσεων είχαμε δεσμευτεί για, να πληρώσουμε για το 2011 5,4 δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι το 2007. Δηλαδή 15,7% περισσότερο από ό,τι το 2007 για το 2011. Αυτά για την ανάληψη υποχρεώσεων. Στις πληρωμές η κατάσταση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Το 2011 θα πληρώσουμε κατά 27,8% περισσότερο από ό,τι το 2007. 7 δισεκατομμύρια περισσότερα. Γιατί τα ταμεία της συνοχής ε, κερδίζουν το χαμένο έδαφος. Και παρόλα αυτή η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από την περίοδο 2006-2007. Και αυτό είναι το καθήκον της Επιτροπή μας, να διερευνήσει γιατί ορισμένες χώρες, και κοιτάξτε τον πίνακα που σας έδωσα, γιατί ορισμένες χώρες έχουν μείνει πίσω. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν προβλέπει αρκετά κονδύλια. Γιατί σε άλλες πολιτικές έχουμε πολύ μικρότερες πληρωμές, λιγότερες πληρωμές για το 2011 από ό,τι στο 2010. Ενώ στην περιφερειακή πολιτική έχουν αυξηθεί αλλά η χρησιμοποίηση των κονδύλιων στις διάφορες χώρες δεν είναι ικανοποιητική. Ευχαριστώ, Λάμπερτ Βανίστερο. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε χρόνο, στα πλαίσια της προετοιμασίας του προϋπολογισμού, βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να προσέχουμε να πάει καλά η συζήτησή μας με το Συμβούλιο. Να παραμείνουν τα συμφωνημένα πλαίσια οι αναλογίες, τα σχήματα πάνω στα οποία έχουμε αποφασίσει να δουλέψουμε να μην αλλάζουν. Όμως, στηρίζουμε τον εισηγητή απόλυτα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα. Πριν από δύο μήνες, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είδαμε ότι συζητήθηκε η πολιτική συνοχή, τα αποτελέσματά της, ότι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια καλή στιγμή, θετική. Μην κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα από ό,τι είναι, από την πλευρά μας λοιπόν. Ένα πράγμα θέλω εδώ να υπογραμμίσω. Μπορεί να φαίνεται ε, ασήμαντο, αλλά μερικές φορές τις λεπτομέρειες είναι η σημασία. Λοιπόν, η Επιτροπή μας όσον αφορά την προετοιμασία Συνηθίζουμε μαζί εδώ να κοιτάμε ποια είναι τα σημεία που πιστεύουμε ότι αποτελούν μια νέα πολιτική που θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε και άλλα που βλέπουμε πώς προχωράει η πολιτική μας. Όμως ο σχεδιασμός που έχουμε προβλέψει δεν ε, ικανοποιεί τα σχέδιά μας αυτά. Είναι πράγματα που συζητάει η Επιτροπή Προπολογισμών χωρί να έχουμε εμεί συζητήσει προηγουμένω. Δεν θα έπρεπε να τα είχαμε δει και εμεί, να τα είχαμε βάλει στην ημερήσια διάταξη πριν. Εν πάση περιπτώσει. Πάντω, το περιεχόμενο, για το περιεχόμενο πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε τρία σχέδια. Και αν δείτε τώρα εδώ, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Για το έρασμο που είχαμε συμφωνήσει, Πού το. Γιατί. Γιατί δεν έχουμε τις πληροφορίες που θα έπρεπε. Έπειτα εμεί ως ομάδα, ως ΕΛΚΑ, θέλουμε κάτι για τις πόλεις και για την Ήπεθρο. Δεν πρέπει να είναι δύο πράγματα τα οποία να πηγαίνουν παράλληλα, πρέπει και τα δύο να τα δούμε. Αυτές είναι προτάσεις που υπάρχουν, ad hoc βέβαια, και θα έπρεπε να προωθηθούν. Αλλά τώρα είναι αργά. Ως Περιφερειακή ε, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μείνει κάπως πίσω. Είναι πολύ αργά για να τα βάλουμε τώρα. Ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν προτάσεις. Οπότε πρέπει να ξαναδούμε τις διαδικασίες. Τι να κάνουμε, κάθε ομάδα να προτείνει κάτι στην Επιτροπή μας, αλλά θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και να προβλέπεται ένας ολόκληρος κατάλογος και μετά να δούμε τι νέες πρωτοβουλίες θέλουμε να υποστηρίξουμε. Έχω μιλήσει για ένα New Pilot Urban πρόγραμμα. Να δούμε τις διαδικασίες λοιπόν για να μπορούμε να τα συμπεριλαμβάνουμε αυτά. Η Πρόεδρος. Κάπως σύντομα θέλω να σας εξηγήσω για αυτά που είπε τώρα ο Λαμπέρ. Θα θυμόσαστε ότι συζητήσαμε στην Επιτροπή μας την προηγούμενη, την προπροηγούμενη προφορά, ε, φορά ήταν για τη διαδικασία τη φετινή. Και έχουμε κάνει προπαρασκευαστική εργασία. Είχαμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει να μας παρουσιάσει την κατάσταση πραγμάτων, της, ε, την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τα πειραματικά προγράμματα. Τα συζητήσαμε στην Επιτροπή μας. Και τώρα όντως υπήρξε αυτή η άτυπη ευκαιρία που μας δίνει η νέα ρύθμιση, οι πολιτικές ομάδες να μπορούν επίσημα να παρουσιάσουν τα προγράμματα εκείνα τα οποία θα ήθελαν να συμπεριληφθούν και να αξιολογηθούν στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά επίσημα να μπουν στην διαδικασία της Επιτροπής μας για να συμπεριληφθούν μετά το καλοκαίρι στον προπολογισμό. Για τα πειραματικά προγράμματα όντως έχει παραταθεί η προθεσμία και έχει γίνει 21 Ιουνίου, έτσι δεν είναι. 4 Ιουνίου ήταν ε, η προθεσμία που έθεσε η Επιτροπή Προπολογισμών. Για εξηγήστε μας η γραμματεία. Η Επιτροπή Προπολογισμών έθεσε προθεσμία για προτάσεις από τις διάφορες επιτροπές την 4η Ιουνίου, ώστε να στείλει μια ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 7 Ιουνίου. Πήραμε λοιπόν πέντε πειραματικά προγράμματα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και, θα... και προωθούνται από τη Γραμματεία μέσα στις προθεσμίες στην Επιτροπή Προπολογισμών. Πρόκειται για κάτι προπαρασκευαστικό, όπως είπε και ο κύριος Σούριον για να πούμε στην Κομισιόν, να, κάποιες ιδέες που έχουμε, κοιτάξτε κατά πόσο μπορούν να προχωρήσουν ή όχι. Η προθεσμία τώρα, η τελική και οριστική προθεσμία για πειραματικά προγράμματα για οτιδήποτε τροποποίησης, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο. Αλλά αν μιλάμε τώρα για την γνωμοδότηση τον Ιούλιο, αν μπορούμε να έχουμε κάτι μέχρι τις 21 Ιουνίου, εμείς στη Γραμματεία, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πράγματι τον Ιούλιο. Εκεί κολλάει η προθεσμία της 21ης Ιουνίου. Θέλω να πω ότι ακόμα μπορείτε να προτείνετε προγράμματα όλες οι πολιτικές ομάδες. Έχουμε πάρει από τους φιλελεύθερους, από το ΕΛΚ, δύο από τους πράσινους, τίποτα από τους σοσιαλιστές, αλλά μπορείτε ακόμα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, η τελική αξιολόγηση θα γίνει ακόμα από την Επιτροπή. Έχουμε συζητήσει κάποια πειραματικά προγράμματα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα εσείς στις πολιτικές ομάδες μπορείτε ακόμα να δουλέψετε και θα επανέλθουμε για να αποφασίσουμε ως Επιτροπή Περιφερειακών ε, Υποθέσεων τις προτεραιότητές μας. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Η Κωνσταντ Σακρέλη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον συγκητή εκφράσω την ε, ευχή να καταφέρει τόσο ως προς τις ε, πιστώσεις χρειάζεται, όσο και προς, προς τις πληρωμές να έχει τα ποσά τα οποία χρειάζεται. Δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνουν οι συνθήκες που όντως αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, δύσκολες συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τη δυνατότητα στην τελική ψηφοφορία της πρώτης περίοδου του 2006 να πιέσουμε και να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των ταμείων συνοχής. Ο εισηγητής είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων τα οποία δεν έχουν πράγματι αξιοποιηθεί, ότι πράγματι δεν έχουν καταβληθεί. Είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε εδώ και πολλά χρόνια. Το Συμβούλιο όμως πάντοτε βρέθηκε απέναντί μας, πάντοτε φρέναρε αυτές τις ε, προσπάθειες. Αλλά εμείς είμαστε κοινοβούλιο δεν είμαστε συμβούλιο. Έχουμε διαφορετικά συμφέροντα σε τελευταία ανάλυση από το Κοινοβούλιο και εμεί, ειδικά από την ομάδα μου, έχουμε κάθε συμφέρον και βούληση να ενισχύσουμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή τη μεταφορά των κονδυλίων που δεν έχουν απορροφηθεί. Για τα πιλωτικά σχέδια, εδώ και πολλά πολλά χρόνια εγώ συμμετέχω είτε ως αναπληρωματικό του τακτικό μέλος στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και πρέπει να πω ότι όντω δεν κατατέθηκαν πιλωτικά σχέδια εφέτος. Θα πρέπει λοιπόν ως Επιτροπή να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε εάν μπορούμε να έχουμε πέντε πιλωτικά σχέδια εμεί ω Επιτροπή των Προπολογισμών. Τη διαδικασία τη γνωρίζετε βέβαια. Η διαδικασία των προπολογισμών δεν αλλάζει κατ' ουσίαν με τη νέα συνθήκη. Και άρα ίσω θα πρέπει να δούμε στα πιλωτικά σχέδια, που στα τελευταία ανάλυση πρόκειται για μικρά κονδύλια, όχι τόσο μεγάλα. Ίσως θα ήταν καλό όμως να κάτσουμε, να συζητήσουμε με το brainstorming όπως λέμε, μερικές ώρες να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε την έμφαση στα πιλωτικά σχέδια. Και πρέπει πιστεύω με επικριτικό βλέμμα να διαλέξουμε πέντε πιλωτικά σχέδια για τα οποία θα έχουμε εγγυημένη υποστήριξη από τον προϋπολογισμό. Έχει γίνει συζήτηση και για το κατά πόσον λειτουργεί το πρόγραμμα Εράσμους, το κατά πόσον η στήριξη σε αυτό ή σε άλλα προγράμματα πηγαίνει προς το στόχο που είχε αρχικά σχεδιαστεί και εάν θα πρέπει να διατηρηθούν. Όλα αυτά μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε λοιπόν. Το μικρό περιθώριο που αναφέρθηκε, εγώ θεωρώ ότι είναι κατανοητό για σε τελευταία ανάλυση έχουμε να κάνουμε με περιορισμένο περιθώριο χειρισμών στην ε, προκειμένη περίπτωση και δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση τώρα. Ίσως με τις συζητήσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχή θα ήταν σκόπιμο να συζητήσουμε αν μπορούμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία και σε μελλοντικέ περιόδους κρίσεως να έχουμε περισσότερη, ε, ταχύτερη μάλλον δυνατότητα αντίδρασης. Προς το παρόν όμως δεν νομίζω ότι μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό το ζήτημα των περιθωριών. Κατά τα άλλα βέβαια η ομάδα μου σας υποστηρίζει και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή και στεναρή παρουσία της Επιτροπής των Περιφερειών στην υπόθεση αυτού του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ρίκα Ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες Όμω θέλω να αναφερθώ σε ένα πιο ειδικό θέμα, σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να μιλήσω για τις περιοχές που χρηματοδοτούνται όσον αφορά τη Βαλτική θάλασσα. Όταν ετοιμάσαμε τη στρατηγική και κοιτάξαμε τις τροπολογίες της ΑΦΕΤ, διαπιστώσαμε ότι είχαμε προτάσεις για μια ξεχωριστή γραμμή στον προπολογισμό όσον αφορά την Βαλτική ε, θάλασσα που θα πήγαινε από το 4 στο 1β, από το τίτλο 4 στο 1β που είναι για την πολιτική συνοχή. Εγώ πιστεύω ότι και εδώ ως ε, Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί αν αρχίζουμε και χρηματοδοτούμε ε, με ξεχωριστές γραμμές στον προπολογισμό τέτοια θέματα τότε αυτό τι σημαίνει στην πράξη για το Ταμείο Συνοχής και για την πολιτική μας συνοχής. Η Επιτροπή μας δεν το έχει συζητήσει αυτό το θέμα, ενώ θα έπρεπε. Και ως ε, αναπληρώτρια στην Επιτροπή Προπολογισμών ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη πίεση εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να το συζητήσουμε ώστε τέτοιες αποφάσεις να μην ε, έρχονται σαν, έκπληξη, σαν σε εμά από άλλε επιτροπέ. Άλλο σύντομα παρακαλώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εισηγητή για την ποιότητα της εργασίας, λέει η κυρία Κόνα. Η κυρία Κόνα. Για την ε, πολιτική συνοχή λοιπόν μιλάμε τώρα και διαπιστώνουμε ότι το ποστό χρήσης των κονδυλίων δεν είναι ικανοποιητικό. Έχω την τάση να σκέφτομαι ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι αρκετά ελιστική. Και θα σας δείξω γιατί το εννοώ, θα σας το πω. Λοιπόν, η σημερινή πολιτική συνοχής ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2007. Τέθηκε σε εφαρμογή και αποφασίστηκαν οι διάφοροι προσανατολισμοί το 2005. Μέσα σε μια συγκυρία που ήταν εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Η οικονομική κρίση λοιπόν που μας πλήττει σήμερα ήταν κάτι που κανείς δεν είχε φανταστεί το 2005 τότε που καθορίστηκαν οι μεγάλοι προσανατολισμοί της πολιτικής συνοχής. Κανείς δεν τα είχε φανταστεί όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει κανείς δεν τα είχε φανταστεί έτσι όπως έγιναν στην πραγματικότητα με τη βία με την οποία μας έφτασαν και έπληξαν τα κράτη και τις επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει την πολιτική συνοχής είναι η έλλειψη ελαστικότητάς τη και σύνδεσή της με τη σημερινή συγκυρία. Και γι' αυτό και η χρήση των κονδυλίων είναι τόσο ανεπαρκής. Και φοβάμαι ειλικρινά ότι θα έχουμε δυσκολίες να κερδίσουμε έδαφος και να καλύψουμε τη διαφορά μέσα στην προθεσμία που έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κρέλ για το ότι πρέπει να προσπαθήσουμε οι χώρες να κρατήσουν τα ποσά που δεν χρησιμοποίησαν κάποιες περιφέρειες σε εθνικό επίπεδο. Τι εννοώ, μια περιφέρεια η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο του φακέλου που έχει στη διάθεσή της, το χρημάτο που έχει στη διάθεσή της, να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει το κράτος για μια άλλη περιφέρεια. Τέλος. Η ιδέα ενός εράσμους των τοπικά εκλεγμένων για μένα είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Γιατί έτσι οι τοπικά εκλεγμένοι, οι τοπικοί άρχοντες και οι τοπικοί παράγοντες θα μπορούσαν έτσι να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να γίνονται καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί για να επωφεληθούν από την πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λάσλο, θέλεις ένα λεπτό για να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους που πήραν το λόγο εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω όλα αυτά στο τελικό μου σχέδιο. Τώρα, μια που δεν έχουμε χρόνο, το μόνο που θα πω είναι τα εξή. Η κύρια φιλοδοξία μας θα πρέπει να είναι να στηρίξουμε τη θέση της Επιτροπής. Η Επιτροπή έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για την περιφερειακή πολιτική και ο καυγάς θα γίνει ανάμεσα στο Συμβούλιο και εμάς. Εμείς στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το βασικό λοιπόν, η κύρια φιλοδοξία μας για να συμπεριλάβουμε ό,τι θέλουμε. Το δεύτερο είναι τα πειραματικά προγράμματα που επίσης θέλουμε να στηρίξουμε. Γι' αυτό που είναι εδώ, δεν είναι πια εδώ, διαφωνώ λιγάκι με τη θέση των σοσιαλιστών, γιατί σε αυτό το στάδιο καλό είναι να έχουμε έναν μακρύ κατάλογο. Και αν ο μακρύς κατάλογος αυτός στηριχτεί από μια ειδική επιτροπή όπως είναι η δικιά μας, που ειδικεύεται στην περιφερειακή πολιτική, τότε το πρώτο κομμάτι θα ενισχυθεί. Αναφίβολα, έτσι. Είναι ψυχολογικό αυτό το θέμα. Αυτό θα γίνει στην Επιτροπή Προπολογισμών. Και αυτό θα βγει από τις διαπραγματεύσεις. Τώρα για τα συγκεκριμένα πειραματικά προγράμματα, ωραίες ιδέες, τις θέλει το Κοινοβούλιο, όχι όμως απαραίτητα και η Επιτροπή, η οποία υπόσχεται ότι θα αξιολογήσει, ότι θα μας στείλει μελέτη κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι στον τομέα αυτό θα πετύχουμε. Δεν νομίζω. Η ιδέα είναι καλή. Εγώ θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες και για τις μικροπιστώσεις ως πειραματικό πρόγραμμα πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά την σχέση που έχει αυτό το πρόγραμμα με τις νέες ε, μικροοικονομικές διευκολύνσεις που ξεκίνησαν φέτος. Γιατί έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι περιττό, εφόσον έχουμε καλύτερα εργαλεία στη διάθεσή μας, περισσότερο ισχυρά όπως είναι οι μικροοικονομικές διευκολύνσεις. Για τις προθεσμίες, ευχαριστούμε για την εξήγηση που μας δώσατε. Είναι ξεκάθαρα. Δύο λόγια τώρα για τη συνθήκη της Λισαβόνας που υποσχέθηκα ε, στην παρουσίασή μου, αλλά ήταν κάτι που έμεινε για το τέλος. Λοιπόν, πολλές φορές λέμε ότι εξαιτία ε, της εθήκης της Λισαβόνας η εξουσία, η δημοσιονομική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί. Αυτό είναι στην επιφάνεια γιατί στην πραγματικότητα έχουμε λιγότερες εξουσίες από ό,τι κατά το παρελθόν. Και γιατί, γιατί όλο το σύστημα έχει φτιαχτεί έτσι ώστε πρέπει να συμφωνούν τα διάφορα όργανα. Και υπάρχει μία μόνο κατάσταση όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει από μόνο του. Υπήρξε συμφωνία στην συνδιαλλαγή και το Συμβούλιο καταψήφισε Μόνο σε τέτοια περίπτωση μπορούμε εμείς να ψηφίσουμε όπως θέλουμε. Είναι ρεαλιστικό ο πρόεδρος και όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνούν μαζί μας και μετά να προχωράμε και να καταψηφίζουν τη συμφωνία. Δεν ναι, είναι ρεαλιστικό. Οπότε πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις διαπραγματεύσεις κάθε φορά. Πρέπει να έχουμε καλές συμφωνίες και ισχυρές ε, κόκκινες γραμμές, δυνατά όρια. Να ξέρουμε πού σταματάμε. Αν πούμε όχι, όλο το πακέτο πάει πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να υποβάλουν νέα πρόταση. Και μετά πάμε στα δεκατημόρια. Λοιπόν, προσοχή εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό. Η Προεδρία όμως θέλει να προχωρήσει και το θέλει τον προπολογισμό. Αυτό είναι, αν θέλετε, το σημείο διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε τόσο ισχυρέ εξουσίε όπως κατά το παρελθόν. Γιατί παλιά λέγαμε ορίστε, αυτό είναι το όριο πληρωμών και κάτω από αυτό το επίπεδο μπορούμε να αποφασίσουμε για την κάθε γραμμή από μόνοι μας για τις μη υποχρεωτικέ δαπάνες. Δεν υπάρχει δεύτερη ανάγνωση εκτός από το ναι ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ Λάσλο. Και να υπενθυμίσω στους συναδέλφους για τα πιλωτικά σχέδια ότι εάν τυχόν υπάρχουν πολιτικές ομάδες που ακόμη θα ήθελαν να υποβάλουν κάποιες προτάσεις, παρακαλώ τώρα, τον Ιούνιο, έχουμε και πιο πολύ χρόνο σε τούτου για να προετοιμάσουμε τις αποφάσεις και τις για τις προτεραιότητες μας που θα πρέπει να είναι έτοιμες για την τροποποίηση του προϋπολογισμού προς τα τέλη Αυγούστου μάλλον ή Σεπτεμβρίου. Αλλά τις προτεραιότητες πρέπει να τις έχουμε έτοιμες για τον Ιούλιο. Και προχωρώ στο τελευταίο σημείο της ημερησίας μας διάταξης, που είναι η συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας για συζήτηση με αλφαβητική σειρά ο κύριος Τζον Μπάχτλερ, καθηγητής των Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, τον κύριο Ζων Σαρ Λεγκέ, πρώην αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ζωμαρή Ρουσό, ε, προεθνικό επιρρογνώμονα της Γενικής Διεθνής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Γιάζεκ Ξλάχτα, καθηγητή Οικονομικής Σχολής της Βαρσοβίας. Παρακαλώ τώρα τους επιρρογνώμονες μας να έρθουν εδώ να μας μιλήσουν με τη σειρά που θα επιλέξετε εσείς βεβαίως ε, για τα σημαντικά θέματα. Φυσικά μπορέσετε να ακούσετε και τις σημερινές μας συζητήσει σήμερα, Εξού μπορείτε από αυτά να αντλήσετε ποια είναι τα σημαντικά για το μέλλον της πολιτικής μας ε, από το 2013 και μετά και μετά μπορούμε να προβούμε σε ανταλλαγέ απόψεων. Ε, κύριε Μπάχτλερ, παρακαλώ. Uh, good morning. Um... Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, το όνομά μου είναι Τζον Μπάχτλερ από το Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών, το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών. Μου στήθηκε να μιλήσω για πέντε περίπου λεπτά και γι' αυτό θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες σύντομες σκέψεις για το πού όσο έχει προχωρήσει η συζήτηση περί χάραξη πολιτικής στην περιφερειακή πολιτική και να επισημάνω ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη πτυχή που είναι η αποδοτικότητα της περιφερειακής πολιτικής. βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια θεμελιώδη ζητήματα ως προς το μέλλον της πολιτικής που προκύπτουν. Μπορούμε να πούμε παραδείγματι, να κοιτάξουμε πρώτα ποιο είναι το κοινό πεδίο, όπως θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, τομείς ε, στους οποίους ε, εξασφαλίζεται ευρύτερα συμφωνία. Πρώτον, ε, είναι αναγκαίο να είναι πιο στοχευμένη η πολιτική, να περιοριστεί ενδεχομένω σε πιο περιορισμένο αριθμό, σε πιο μικρό αριθμό προτεραιοτήτων, έρευνα, καινοτομία, οικονομία χαμηλής εκπομπές ε, ε, άνθρακα. Ναι, δεύτερον, πρέπει να είναι πιο ορατή και ορατά τα αποτελέσματά της. Πολλές είναι οι προτάσεις που ακούστηκαν για την υπαγωγή σε όρους, για τις δαπάνες, καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερα ορόσημα. Τρίτον, πολλές από τις παρεμβάσεις υποστηρίζουν περισσότερη στρατηγική συνοχή, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, διαρθρωτικών πολιτικών, μεταξύ των διαρθρωτικών πολιτικών σε άλλους τομείς, και με άλλους τομείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής δηλαδή. Και επίσης θα πρέπει να εξορθολογιστεί ο δημοσιονομικός έλεγχος και οι προϋποθέσεις ελέγχου. Δηλαδή να μην υποβαθμιστεί η αυστηρότητα των ε, κανόνων, αλλά να εξορθολογιστεί ο τρόπος εφαρμογής τους. Τέταρτον, ανάγκη και πάλι για απλουστευσή της γραφειοκρατίας, για κατάρριση γραφειοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό κάθε συζήτηση που έχει γίνει για μεταρρύθμιση τα τελευταία 20 χρόνια και επίσης Γενικά συμφωνία υπάρχει ότι χρειάζεται προσθερή ε, έμφαση να δοθεί στην εδαφική συνεργασία. Σημαντικές όμως είναι και οι αποκλήσεις απόψεων που, εκφράζονται μέσα από το δημόσιο διάλογο. Κύριο σημείο απόκληση. είναι ποιος είναι ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει μια τέτοια πολιτική και ποια είναι η ιδιαίτερη κάλυψή της. Θα πρέπει να εκτείνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πρέπει να περιοριστεί στη στήριξη των πιο φτωχών. Πρέπει να είναι ένας κύριος τομέας ε, πρωταρχικός δηλαδή ή δευτερογενής μόνο, συμπληρωματικά δηλαδή να δρά. Επίσης, διαπιστεύονται κάποιες αποκλήσει απόψεων ω προς τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών πολιτικών Φερρυπίν, Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων στο σύνολό του, αφενό και περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη αφετέρου. Επίση, βλέπουμε και την ε, διαφορετική ε, έμφαση που δίνεται ως προς την ε, συμμετοχή της τοπικής διακυβέρνησης, δηλαδή το κατά πόσον θα πρέπει η εφαρμογή αυτή της, της πολιτικής να είναι κεντρική ή αποκεντρωμένη. Μετά τις ε, σύντομες αυτές παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε κάποιους βασικούς τομείς όπου έχουμε συμφωνία, δηλαδή και όπου εκφράζεται η ανάγκη καλύτερη και πιο ορατή επίδοση των επιδόσεων. Νομίζω ότι ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής που έκανε την αξιολόγηση πολιτικής ε, βοήθησε ιδιαίτερα ε, τις διαπιστώσεις και μάλλον είχατε και τη σχετική παρουσίαση. Πάντως ε, θα πρέπει να δούμε τι προκύπτει από τις διάφορες αξιολογήσεις της πολιτικής και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα ότι φέρνει σημαντικό, σημαντικά αποτελέσματα η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική συνοχής και ως προς την ανάπτυξη του ΑΕΠ και σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης, της απασχολησιμότητας, ιδιαίτερα, προς την ενίσχυση, ιδιαίτερα στον τομέα της ενίσχυση των επιχειρήσεων, τη μείωση των περιφερειακών διαφορών και και επίσης ε, και διοικητική ε, διοικητικές αλλαγές οι οποίες αποτελούν λίγο πολύ ε, την αντανάκλαση των αλλαγών σε, σε κοινοτικό επίπεδο πάνω στο εθνικό επίπεδο. Δηλαδή βελτιώνεται και σε εθνικό επίπεδο η διοίκηση. Ε, φυσικά υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ διαφόρων περιοχών, ε, περιφερειών, μέσα στο ίδιο κράτο ακόμη. Αυτό είναι δεδομένο, ναι, αλλά συνεχίζονται και κάποια θεσμικά προβλήματα τα οποία αποδυναμώνουν την απόδοση μιας καλής πολιτικής συνοχής. Φερρυπίν διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αναλυτική βάση για το σχεδιασμό προγραμμάτων και κοινοτομίας. Διαπιστώνουμε ότι δεν είναι επαρκής η στρατηγική συνοχή μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Φαίνεται ότι υπολοιπόμεθα στην εκτέλεση των ιδεών, δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός ε, στην εφαρμογή, στην υλοποίηση της ε, πολιτικής. Υπάρχουν ε, επίσης αδυναμίες ως προς την χορήγηση των κονδυλίων και παρά τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί δεν είναι πολλές φορές ικανά τα συστήματα να προσφέρουν επαρκείς και έγκαιρες πληροφορίες παρότι είναι αρκετά δεδομένη πλέον η διαδικασία της αξιολόγησης πάλι ποικίλει η ποιότητα των αποτελεσμάτων και ο χρονισμός τους. Τα προβλήματα φυσικά δεν εμφανίζονται ομοιόμορφα σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. Υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα καλών πρακτικών, βέλτιστων πρακτικών στις περιοχές αυτές, όπως υπάρχουν και παραδείγματα αδυναμιών και ε, ε, ελλείψεων. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχουν αυτοί οι θεσμικοί περιορισμοί που είχαμε δει ήδη στην στο προηγούμενο διάλογο για την μεταρρύθμιση και τη, στη δεκαετία του 2000 αρχές αλλά και στη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει με σοβαρότητα να εξεταστούν ε, ω ε, τμήμα του τωρινού δημόσιου διαλόγου. Θα πρέπει παραδείγματι μαζί να επανεξεταστεί το σύστημα του, ε, της πολυεπίπεδης διαχείρισης που είναι πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα αποτελεί και πηγή κάποιων δυσκολιών ή ελλείψεων. Είναι κάτι το οποίο καταγράφει και η έκθεση Μπάρκα στην έκθεσή τη, το σύστημα δηλαδή των, ε, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ένα από τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού στη λειτουργία του συστήματος πολυ, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι το να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την αποτελεσματική και σωστή διάθεση των κονδυλίων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα, ε, στο οποίο θα επανέλθω σε λίγο. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η στρατηγική συνοχή της παρέμβασης. Ήδη αναφέρθηκα σε κάποιες προκλήσεις που εμφανίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο υπάρχουν προκλήσεις και για τα κράτη-μέλη. Προκλήσεις που έχουν σαν συνέπεια ή μάλλον που δεν ε, αντιμετωπίσουν σωστά γιατί δεν υπάρχει όραμα ω προ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ε, προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν στρατηγικά, στα στρατηγικά έγγραφα αλλά όχι στην πράξη. Σημαντικά ζητήματα επίση είναι αυτά ε, τη ικανότητα ε, των θεσμών να δράσουν σε δεδομένε καταστάσει. Αυτό ήδη έχει επισημανθεί πιστεύω. Και ταυτόχρονα σαφές καθίσει το γεγονός ότι ναι, μερικές φορές υπάρχει σωστή διαχείριση των ε, παρεμβάσεων, διατίθεται τα χρήματα, υπάρχει λογοδοσία ως προς το που διατίθενται, αλλά λείπει πάντα μία συνέπεια, συνέπεια όραμα ή συνοχή ως προς την προσέγγιση. Εν τέλει θα ήθελα να επισημάνω την έλλειψη λογοδοσίας που χαρακτηρίζει την ε, πολιτική. Αυτό οφείλεται σε στα προγράμματα ίσως, δηλαδή εντοπίζεται στο επίπεδο του προγράμματος. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή υποχρέωση λογοδοσίας του γιατί δεν επετέχθησαν οι στόχοι, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ επανέρχομαι στη σύσταση της έκθεσης Μάρκερ για το για την ανάπτυξη ενός φόρουμ υψηλού επίπεδου που θα συζητήσει και θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα επιτεύγματα της πολιτικής να τα συζητούν τα κράτη-μέλη και να εξασφαλίζουν μια ε, κάποια ε, λογοδοσία. Σας ευχαριστούμε. Ε, Ο κύριος Λέγκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τη μελλοντική περίοδο που είναι η κεντρική περίοδος και το αντικείμενο συζήτησης ε, και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, ε, διαρωτόμαστε κατά πόσο η πολιτική συνοχή είναι, εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Η συζήτηση γίνεται για το κατά πόσο όντω πρόκειται για προστιθέμενη αξία ή όχι. Ποιε θα ήταν οι προποθέσει. Αυτή είναι βέβαια και η αιώνια συζήτηση που γίνεται εδώ και 20 χρόνια για την πολιτική συνοχή. Νομίζω ότι το πρώτο θέμα που πρέπει να επενθυμίσουμε για να μην υπάρχει αμφισημία για το τι είναι πολιτική συνοχή είναι να υπενθυμίσουμε ότι πρώτα απ' όλα είναι μια διαρθρωτική δράση μακροπρόθεσμη η πολιτική συνοχή. Δεν είναι συγκυριακή πολιτική. Για τελειώσει η πολιτική συνοχή δεν έχει νόημα. Τρίτον, δεν είναι μια πολιτική εσόδων. Στόχος της δεν είναι κατά κύριο λόγο να αποτελέσει ένα εργαλείο για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην κοινωνική ένταξη. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, γιατί αλλιώ υπάρχουν παρεξηγήσεις όσον αφορά το τι μπορεί να προσφέρει η πολιτική συνοχή. Δεύτερον, πρέπει να υπενθυμίσουμε, και εμείς το ξέρουμε αυτό καλά, ότι σε 20 χρόνια η πολιτική αυτή εξελίχθηκε προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτον, επικουρικότητα αυξανόμενη συνεχώς και πλήρης όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων από τις χώρες και τις περιφέρειες. Από την άλλη μεριά όμως είχαμε και μια αύξηση των ελέγχων ε, των κονδυλίων παρόλο που τα κράτη-μέλη έχουν τον κύριο ρόλο, αλλά επειδή η συνθήκη το προβλέπει, η Κομισιόν έχει αποφασιστική σημασία ρόλο για την ε, εκτέλεση των ε, κονδυλίων. Υπό το φως λοιπόν αυτών που υπενθύμησε και που είναι προφανή, μπορούμε στο χρόνο που μου διαθέσατε κυρία Πρόεδρε να αναρωτηθούμε για τα εξής τρία. Πρώτον, το περιφερειακό επίπεδο είναι το κατάλληλο πάντα για την πολιτική συνοχής. Ξέρουμε ότι γίνεται πολιτική συζήτηση σήμερα για αυτό το θέμα. Δεύτερον, η λειτουργία της πολιτικής συνοχής είναι να μειώσει τις διαφορές πάντα πρέπει να συνεχίσει να είναι αυτό. Και τρίτον, που το επενθύμησε και προηγουμένως, η διαχείριση της πολιτικής συνοχής είναι το κύριο στοιχείο σε σχέση με το οποίο πρέπει ενδεχομένω να αλλάξουν τα πράγματα για να έχουμε καλύτερη απόδοση. Το πρώτο θέμα, κατά πόσο το περιφερειακό επίπεδο είναι το κατάλληλο σε σχέση με το εθνικό ή σε σχέση με το κατατομής. Υπάρχει συζήτηση γι' αυτό, συζητιέται. Δύο διαπιστώσει σύντομα, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε για τι πράγμα μιλάμε. Έχουμε 27 μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 προσπαθεί να ανταποκριθεί στη διαπίστωση που λέει ότι οι περισσότερες 55% των περιφερειών από τις 171. Οι περισσότερες λοιπόν έχει ένα επίπεδο ευημερία ΕΠ χαμηλότερο από το όρο Το 55% ε. Περισσότερες από τις μισές. Το χάσμα δηλαδή που υπάρχει και οι συνθήκες ανταγωνισμού στις περιφέρειες αυτές, είτε είναι κάτω από το 5% ή είναι ανάμεσα στο 5% και το 100%, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Άρα το σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας ως επιτοπλίστου αντιμετωπίζει δυσκολίε ανταγωνισμού και ανάπτυξης. Δεύτερον, για τις περιφέρειες οι οποίες είναι λίγο πάνω από τον κοινοτικό μεσόρο, 104 περιφέρειες, πάνω από το 1 τρίτο δηλαδή, είναι στην ψαλίδα 100-150%. Και οι ανταγωνιστικές που έχουν ε, τις ίδιες διαφορές όπως έχουμε περίπου στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία είναι ελάχιστες. Είναι 15 περιφέρειες από τις 271. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαφορές που υπάρχουν όχι μόνο στο εσωτερικό, για να λάβουμε υπόψη μας αυτά που λέει η συνθήκη που μιλάει για αρμονική εξέλιξη, αλλά και στα πλαίσια της ε, παγκοσμιοποίησης. Κάτι άλλο που θέλω σύντομα να επενθυμίσω ποια είναι η κατάσταση στις διαφορές ανάπτυξης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τη συγκρίνουμε με τους μεγάλους ανταγωνιστές μας. Της τάξης 1 μέχρι 8, 1 με 2 και μισό στην Αμερική και 1 με 2 στην Ιαπωνία. Η πολιτική συζήτηση λοιπόν που γίνεται σήμερα για τις ανακλάδο πολιτικές είναι το κύριο θέμα και η πόλη συγκέντρωση είναι στον αντίποδα της στρατηγικής του 2020 που ετοιμάζουμε. Αυτό θέλω να τα υπενθυμίσω για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Τρίτον, η λειτουργία της πολιτικής συνοχής. Είναι να μειωθούν οι διαφορές που υπάρχουν. Να υπενθυμίσω πρώτον ότι η συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε με το άρθρο 174 τη μείωση των διαφορών με προτεραιότητα στην καθυστέρηση ανάπτυξης, στις ε, βιομηχανικές περιοχές, αγροτικές περιοχές κλπ. Όντω αυτή είναι η αποστολή της πολιτικής συνοχής και δεν υπάρχει κι άλλη. Η συνθήκη της Λισαβόνας ψηφίστηκε πριν από πολύ λίγο χρόνο. Τρίτον, τονίζει το ότι πρέπει στα πλαίσια τα περιφερειακά να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν σε διάφορες περιφέρειες, είτε πρόκειται για αστικές, είτε για αγροτικές, είτε για απόμακρες περιοχές. Άρα παραμένει η έννοια της μείωσης των διαφορών. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχουν δύο πολιτικές που προτείνονται. Εναλλακτικέ. Η μία είναι προτεραιότητα να δοθεί στις πολιτικές ανακλάδο, ανατομέα. Και ποιες θα ήταν οι συνέπειες σε αυτή την περίπτωση. Πρώτον, ενίσχυση αποκλειστικά οικονομικών τομέων που είναι πιο ανταγωνιστικοί και αύξηση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών. Δεύτερη εναλλακτική λύση που συζητιέται είναι να επικεντρώσουμε την πολιτική συνοχή στο εθνικό επίπεδο και όχι στο περιφερειακό επίπεδο. Με τη συνέπεια. Η συνέπεια θα ήταν, και συζητήθηκε πριν εδώ κατά πόσο το ΑΕΠ είναι το σωστό κριτήριο, όχι, η συνέπεια θα ήταν ότι το ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Άρα, μείωση των οικονομικών μέσων. Δεύτερον, αυτό θα σήμαινε ότι η δυνατότητα των περιφερειών να αποτελούν εταίρο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 που τόσο συζητιέται τελευταία, εξαφανίζεται πλήρως. Δεν θα είναι πια ετέρη. Είναι κάτι που θέλουμε. Κατά συνέπεια, η σημερινή αρχιτεκτονική της πολιτικής αυτής ήταν ένα πρόβλημα. Για ποιον όμως. Είναι ένα πρόβλημα για τα κράτη-μέλη, ή για αυτούς που πιστεύουν στην επαναθενικοποίηση μέσω του, της μεθόδου ανοιχτού συντονισμού και χωρίς ευρωπαϊκό προπολογισμό. Για αυτές τις χώρες ή για όσους υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, η λύση είναι απλή. Εξαφανίζεται η πολιτική συνοχής και τον τίνουμε αυτό με μια ευρωπαϊκή δράση χωρίς όμως ευρωπαϊκή ανάμειξη. Η δεύτερη λύση, η αποκλειστική στήριξη των μεγάλων ε, πόλων ανταγωνισμού, είναι μια λύση. Ξέρουμε ότι αυτή η λύση οδηγεί στην αύξηση των διαφορών. Δεν θα είναι ένα με 8, θα είναι πολύ παραπάνω. Και το δικό μας το επίπεδο ανταγωνισμού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, ΗΠΑ για παράδειγμα, θα αυξηθεί. Η τρίτη εναλλακτική που συζητιέται είναι μια πολιτική συνοχή σε εθνικό επίπεδο μόνο. Εξαφανίζεται το περιφερειακό επίπεδο δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση γίνεται ανάμεσα στα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαφανίζεται λοιπόν η εταιρική σχέση με τις περιφέρειες και η ειδική συγχρηματοδότηση. Ο προσανατολισμός που πρέπει να βρούμε είναι πώς θα συνεχίσουμε τη σημερινή αρχιτεκτονική, αλλά λαμβάνοντας υπόψη καλύτερα τις περιφερειακές ανάγκες. Συνεπώς, η προτεραιότητα πρέπει να μείνει στις περιφέρειες που βρίσκονται πιο πίσω, τις περιφέρειες σύγκλησης όπως ονομάζονται. Και δεύτερον, αυτό που σήμερα ονομάζουμε περιφέρειες με ανταγωνιστικές και για την απασχόληση, το είπα και πριν, ναι, αλλά πού βρίσκονται αυτές στην Ευρώπη, σε τεράστιες δυσκολίες απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε η ευρωπαϊκή παρέμβαση δεν έχει προστιθέμενη αξία για αυτές τις περιφέρειες, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η προσπάθεια που γίνεται για δημόσιες επενδύσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μειώνονται. Η λύση λοιπόν θα ήταν η μείωση ή η εξαφάνιση ευρωπαϊκής παρέμβασης. Τρίτον, είναι ξεκάθαρο ότι συζήτηση για ένα μεταβατικό στάδιο για τις χώρες που βγαίνουν από τη σύγκληση και εκείνες που βρίσκονται μακριά, πρέπει να γίνει πολύ σοβαρά. Η οικονομική η ειδική παρέμβαση θα είναι κάτι αναγκαίο. Κυρίως μάλιστα μετά από αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, η συνέπεια της οικονομικής κρίσης δεν είναι οικονομικά σήμερα στη δυνατότητα παρέμβασης. Έπειτα το 2011 και 2012 τότε θα έχουμε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης και σε κοινωνικό επίπεδο. Άρα το ζήτημα που και το 2014 είναι πέρα από μια ταχεία αντίδραση που θέλουμε θα έχουμε ένα καλύτερο οικονομικό μέσο και δεν μιλάω τώρα για τα καθαρά υπόλοιπα. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστούν καλύτερα οι ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο, για την κάθε περιφέρεια. Για να λάβουμε υπόψη μας στις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα, που συγκεντρώνουν περιοχές ε, κοινωνική, κοινωνικού αποκλεισμού. Έπειτα να δούμε τις μεσαίες πόλεις, που είναι και οι περισσότερες και για τις αλλαγές στη γεωργία και για οικονομικές και βιομηχανικές αλλαγές και να δούμε και την διασύνδεση μεταξύ περιφερειών. Εκεί είναι που έχουμε να κάνουμε με την εδαφική συνοχή. Αλλιώς κατακαιρματίζεται το θέμα της ένταξης. Και θα τελειώσω τώρα με το εξή, κυρία Πρόεδρε. Η διαχείριση της πολιτικής συνοχής είναι πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα, όπως πάντα, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μην μιλάμε ξύλινη γλώσσα εδώ που βρισκόμαστε και έχω την ευκαιρία συχνά να έρθω εδώ. Πιστεύω ότι επί της ουσίας η σημαντική συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και για την διαχείρισή της είναι το εξής. Η συζήτηση για την επικουρικότητα έτσι όπως έχει προχωρήσει μέχρι τώρα είναι κάτι ικανοποιητικό, είναι ρεαλιστικό. Όχι, κατά τη γνώμη μου. Γιατί η συμφωνία για επικουρικότητα μέσω των κυβερνήσεων, προγραμματισμό, επιλογή προτεραιοτήτων, συγχρηματοδότηση και αποτελέσματα που μέχρι τώρα έχουν αρνηθεί οι περιφέρειε να μιλάνε για αποτελέσματα και κρύβονται πίσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα κάνει αυτά και α κάνει καλά με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε σοβαρή συζήτηση και να δώσουμε την ευθύνη στι περιφέρειε για του στόχου του. Και ο Πασκλετρό είπε πολύ καλά πριν ότι χρειάζεται διάγνωση. Και η διάγνωση δεν γίνεται πάντα σωστά από τι περιφέρειε. Άρα, ούτε και οι προτεραιότητε που επιλέγονται είναι πάντα οι και τρίτον, μέχρι τώρα οι χώρε μα σε εθνικό επίπεδο να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Και η περιφέρειά μας δεν θέλησαν ποτέ να κάνουν συζήτηση για τα αποτελέσματα. Οπότε το κεντρικό ζήτημα για την διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων, είναι να δούμε και τα αποτελέσματα. Και έτσι να υπάρχει μια προαίρεση. Να το συζητήσουμε αυτό. Υπό ποιου όρους Μπορεί να μην αρέσει σε κανένα, να μην ακούγεται καλά, αλλά μετά την απόφαση της 9 η Μαΐου από τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων βλέπουμε ότι η δημοσιονομική συζήτηση θα αλλάξει φύση και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι σε αυτή τη συζήτηση υπαρκτός. Οπότε, το θέμα των προϋποθέσεων ή θα είναι επικίνδυνο να το συζητήσουμε ή θα μιλήσουμε μακροοικονομικά. Φοβάμαι ότι θα καταργηθεί ο περιφερειακός προγραμματισμός γιατί δεν θα χρειάζεται. Θα φτιάχνουμε μια επιταγή για το ένα ή το άλλο κράτος μέλος και το ΕΚΟΦΗΝ, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ θα αποφασίζει ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία όμως δεν θα έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα την αναπτυξιακή των περιφερειών. Θα εξαφανιστεί δηλαδή η διακυβέρνηση που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής αυτής. Ακόμα και αν είναι δύσκολο να δούμε τη σχέση των τοπικών παραγόντων με το μέλλον. Το θέμα αυτό λοιπόν των προϋποθέσεων πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για να εξαρτάται το θέμα αυτό των προϋποθέσεων της χρηματοδότησης από τις ειδικέ ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Και να δούμε πώς θα εκτελείται η πολιτική συνοχής ανάλογα με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Παραδείγματα, χωρίς να είναι εξαντλητικός ο κατάλογος συχνά αποτελεί ψευδέστηση να χρηματοδοτούμε διαφορετικέ επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, ενώ οι ευρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον δεν έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Και αυτό συμβαίνει σε πολλέ χώρες μέλη. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της κοινοτική νομοθεσίας πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση γιατί μόνο τότε μπορεί να είναι αποτελεσματική η επιπλέον χρηματοδότηση που έρχεται από την πολιτική συνοχής. Δεύτερον, πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση ανάμεσα στη διάγνωση που αφορά μια περιφέρεια, που μπορεί να έχει χύψη και τι αιτίε για τι οποίε είναι αυτό το ΑΕΠ 60 ή ξέρω πόσο τη 100. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικέ οι αιτίε στη Γαλαβρία, στην Εστονία ή στο φρανσκοντε συνεπω η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται σοβαρά για τι αιτίε οι οποίε έχουν οδηγήσει σε ένα ΑΕΠ ή σε μια ενεργία χύψη και η περιφέρεια ή το κράτος, ανάλογα με το πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να αρκούνται στο «Α, υπάρχει επικουρικότητα, εμείς ξέρουμε καλύτερα τι χρειάζεται». Όχι. Ή λοιπόν τον άξονα αποτελούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και για το 2006 θα είναι ευρωπαϊκές πολιτικές ο άξονας, οπότε εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και να φτιάξουμε κανόνες ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε και το λογαριασμό, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ποια είναι τα πολιτικά μέσα τώρα που διαθέτουμε, κυρία Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή χρειάζεται και θεσμική συζήτηση, η οποία δεν έχει γίνει επαρκώ. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για δύο προσανατολισμού. Πρώτον, το Συμβούλιο. Δεν συζητάει παρά μόνο όταν φτάνει στι δημοσιονομικέ προοπτικές. Μόνο τότε συζητάει για αυτά τα θέματα. Όπω υπάρχει μια Οικονομική και Πολιτική Επιτροπή, πρέπει να υπάρχει και μια περιφερειακή πολιτική, η οποία να μην έχει σχέση με την ΚΟΚΟΦ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να υπάρχει λοιπόν μια τέτοια επιτροπή, η οποία να συζητά τακτικά, επιμονή μου βάσεως ουσιαστικά, για τις στρατηγικές επιλογές και για τα προγράμματα τα οποία απορρέουν. Να γίνει αυτή η θεσμική πολιτική συζήτηση και το Κοινοβούλιο από την πλευρά του, που συχνά έρχεται σε αντίθεση με την Επιτροπή και με το ελεκτικό Συνέδριο, να λάβει υπόψη το εξή. Η συζήτηση που γίνεται για το ποσοστό σφάλματος είναι μια αιώνια συζήτηση ανάμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών, την Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο. Και γίνεται μια συζήτηση παράλογη για τη δήλωση αξιοπιστία. Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ευθύνη στα κράτη και στι περιφέρειε να είναι πιο υπεύθυνα. Και γιατί να μην σκεφτούμε για παράδειγμα είτε η Επιτροπή, είτε το Κοινοβούλιο, είτε μαζί να καλούν τη μία την άλλη χώρα, ανάλογα με το θεσμικό σύστημα ενδεχομένω στην περιφέρεια, για να έρθει και να εξηγήσει πώ διαχειρίστηκε τα χρήματα. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη διαιτησία εντό αγωγικών για να αποδραματοποιήσει το θέμα. Γιατί αλλιώ η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Γιατί δεν είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση. Θεσμικά είναι υπεύθυνη. Στην πραγματικότητα όμω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τη διαχείριση των προγραμμάτων την έχει η Βαυαρία, το Νορ Παντεκαλέ, η Γάντι, δεν ξέρω ποιο. Πρέπει λοιπόν ε, θεσμικά να ε, αναλάβει ο καθένα τι ευθύνε του. Το θέμα τώρα τη συγκέντρωση. Για την τρέχουσα περίοδο έχουμε 75% για το στόχο 2, 60% για τις περιφέρειες σύγκλησης, είναι μια πρόοδος. Όμως, να είμαστε ειλικρινεί και θα το θυμόμαστε, οι χώρες μας και το Κοινοβούλιο, θυμάμαι, δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό να αποδυναμώσουν τη συγκέντρωση έτσι όπως προβλέπονταν στη Λισαβόνα. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις λοιπόν είναι ένα πάρτα όλα που δεν βοηθάει την προστιθέμενη αξία. Τόσο λοιπόν η Επιτροπή όσο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει για τις προτεραιότητες στρατηγικής 2020 να επικεντρωθούν σε τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, στην ανταγωνιστικότητα που να βασίζεται στην καινοτομία, την έρευνα και τους ανθρώπινους πόρους. Δεύτερον, τις προϋποθέσεις όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη ενέργεια, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. Και τρίτον, προσαρμογή στην οικονομική αναδιάρθρωση και στις συνθήκες κρίσης και στην ανεργία. Αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητες. Όλες οι προτεραιότητες στρατηγικής 2020 είναι καλές, είναι ευθύνη των κρατών μελών για τις χώρες τους, αλλά την ευθύνη της πολιτικής συνοχής για τις προτεραιότητες αυτές είναι κάτι που να είναι πιο αποτετικό. Αλλιώς θα καταλήξουμε στα ίδια αποτελέσματα που καταλήξαμε και με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε, λέει κύριο Σλάχτα. Εγώ θα υιοθετήσω διαφορετικό πρίσμα από τους συναδέλφους και θα πρέπει να εφαρμόσουμε όχι μόνο την προσέγγιση των φίλων της ε, περιφερειακής πολιτικής αλλά λάβουμε υπόψη και τη δικαιολογημένη κριτική αλλά και την άδικη κριτική γιατί και αυτά τα πρίσματα της ανάλυσης είναι ενδιαφέροντα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ορισμένα σημεία. Σημείο πρώτο. Υπερβολικά βραδεία προσαρμογή των ε, δραστηριοτήτων και μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Έχουμε καταρχήν την οικονομία των τόπων και την οικονομία των νόμων. Αν ε, διαβάσουμε προσεκτικά την έκθεση Μπάρκας, θα δούμε ότι η οικονομία των τόπων είναι άριστα σχεδιασμένη. Αλλά η δεύτερη διάσταση δείχνει ότι η εδαφική συνοχή ίσως είναι το καλύτερο, ο καλύτερος τρόπος για την οικονομία των νόμων. Και δεν μιλούμε μόνο για τη σύνδεση των παραδοσιακών υποδομών, αλλά και για τη δικτύωση, το networking, να ξεπεράσουμε τις συνέπειες της ύπαρξης των συνόρων και να προσθέσουμε και κάτι για την ε, καλύτερη μετάδοση από τα βασικά κέντρα. Σημείο 2. Υπερβολικά βραδύ ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η πολιτική συνοχή είναι υπεύθυνη για κάτι τέτοιο. Όχι. Ελάχιστα για να μην πω καθόλου. και υπάρχει πρόβλημα με το πώς θα ε, επιταχύνουμε και πώς θα ενθαρρύνουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες για να αυξήσουμε το δυναμικό ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πρώτη εκδοχή της στρατηγικής του 2020 δεν περιλάμβανε για την πολιτική συνοχή. Την παρέλειψε αρχικά και μόνο μετά από διαβουλεύσει προσθέθηκε και η πολιτική συνοχή, η, η περιφερειακή και τοπική διάσταση. Προσθέθηκαν τεχνικά, τεχνικά μένα, αλλά όχι και στην πραγματικότητα. Το κόστος το είναι υπερβολικό σε σχέση με τα αποτελέσματα, με το όφελος. Οπότε είναι απαραίτητη η απλούστευση, η αποφυγή της επικάλυψης, γιατί υπάρχει τέτοια επικάλυψη. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Επίσης ε, θα πρέπει να περιοριστεί η γραφειοκρατία ε, γιατί αυξάνει το, το κόστος των διατυπώσεων. Θα πρέπει να μειωθεί και το διοικητικό κόστος για τα μικρά κονδύλια. Αυτό αναφέρθηκε πολλές φορές θα πρέπει να βελτιωθεί η διοικητική κουλτούρα σε ό,τι αφορά την εξοικείωση της με τα συστήματα πολιτικής συνοχής. Αυτά τα είπαν και οι συνάδελφοι. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων πολιτικών είναι σημαντικό στοιχείο, γιατί ε, η πολιτική συνοχή και η περιφερειακή πολιτική είναι ένα τμήμα της συνολικής πολιτικής και δεν μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε ποιοτικό συντονισμό και ψηλό συντονισμό αν οι υπόλοιπε πολιτικές υστερούν σε αυτό. Χρειαζόμαστε ενοποιημένα προγράμματα πολιτικής που θα καλύπτουν όλες τις πολιτικές με εδαφικό αντίκτυπο. Αυτό είναι ένα καλό τρόπο για να εξασφαλίσουμε ένα τέτοιο συντονισμό, αλλά τα προβλήματα τη υπαίθρου και τα αναπτυξιακά προβλήματα άλλων περιφερειών δεν αντιμετωπίζονται αρκετά ως προτεραιότητες. Και τα θέματα αυτά είναι πολιτικά, το καταλαβαίνω. Έχουν πολιτική διάσταση, γι' αυτό δεν θέλουμε να επέμβουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές του 2007. Έλλειψη συγκέντρωσης ε, των ε, παρεμβάσεων. Και υπάρχει και το πρόβλημα το κανονιστικό και των διαβουλεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να καταλήξει ένα σύντομο κατάλογο ενώ τα κράτη-μέλη ζητούν ένα μακροσκελή κατάλογο προγραμμάτων και προτεραιοτήτων και στη συνέχεια διαπραγματεύσει μεταξύ τους ε, ε, γίνεται δύσκολη. Γιατί η διάσπαση των προτεραιοτήτων διασπάει και τη χρησιμοποίηση των πόρων. Προτιμώ λοιπόν συγκέντρωση των προτεραιοτήτων και όχι κατακαιρματισμό των προγραμμάτων. Χρειάζεται μία ελάχιστη συγκέντρωση προτάθηκε και η προσέγγιση του ενιαίου ταμείου με χαμηλό επίπεδο συγχρηματοδότησης που δημιούργησε όμως προβλήματα γιατί το software και το hardware της περιφερειακής ανάπτυξης ε, δεν έχει την ίδια πρόοδο σε όλες τις περιφέρειες και δεν υπάρχει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, το ποσοστό απορρόφησης δαπάνη και με ταχύς ρυθμούς, γιατί η απορρόφηση είναι βραδεία. Βέβαια χρησιμοποιούμε διάφορους δείκτες για να καταμετρήσουμε το... τους δείκτες. Ο πρώτος δείκτης είναι αποτελεσματικότητα, ο δεύτερος είναι οι συνέπειες, τα αυτά αποτελέσματα. Χρησιμοποιούμε μόνο τον τρίτο δείκτη. Φυσικά και η παρατήρηση και η επιτήρηση, μάλλον η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι σημαντικές μέθοδοι. Τώρα, παθολογία των επιλέξιμων προγραμμάτων. Φαίνεται αυτό το πρόβλημα δεν αγγίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το πιο ορατό στοιχείο για το κοινό. Γιατί φαίνονται τα αποτελέσματά του και στις περιφέρειες και στις πόλεις. Αν λοιπόν καταφέρουμε ε, να ασκήσουμε πίεση ώστε να χρησιμοποιηθούν αργόριθμοι διαφανών διαδικασιών όταν έχουμε κάπως παράδοξη κατάσταση και να εντοπίζουμε ατασταλείς και να παρεμβαίνουμε πάρα αυτά, αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά μας. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε είναι ότι υπάρχει κάποια ανελαστικότητα. Να χρησιμοποιήσουμε τα αποθεματικά, τα παρατηρητήρια, να κάνουμε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, να αναπτύξουμε μια κουλτούρα της αξιολόγησης, όλα αυτά είναι χρήσιμες συστάσεις. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να τα τονίσουμε και να τα λάβουμε υπόψη κατά το σχεδιασμό του συστήματος και μετά να ελέγχουμε τα επιμέρους σημεία, να δούμε σε πόσα συμφωνούμε και αν συμφωνούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αλλά όπως είπε και ο Ζαν, θα πρέπει να θυμηθούμε και το κληροδότημα του Ντελόρ που συμπεριλήφθηκε και στη συνθήκη. Ενιαίος ρόλος του περιφερειακού επίπεδου στην πολιτική αυτή. Μην ξεχνούμε αυτά που είπε ο Ντελόρ. Και η συνοχή να είναι στόχος της πολιτικής, πανευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της περιφερειακής πολιτικής για την ε, ένταξη, για την ολοκλήρωση, μια πολιτική που θα είναι κοντά στους πολίτες, έμφαση στη δικτύωση και επίση μακροπρόθεσμη διάσταση αυτής της πολιτικής. Αν θέσουμε μια τέτοια σειρά οροσίμων, μπορούμε να φέρουμε τις υποθετές αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Και ο Ζαμαρί Ρουσό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά όμως, γιατί βρίσκομαι Ελπίζω μόνο να με ακούτε καλά, βρίσκομαι δίπλα ακριβώ στο μικρόφωνο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να περιοριστώ στο χρόνο που μας ε, δώσατε. Θα στηριχθώ στην ε, βασική θέση από το draft position, από το ε, σχέδιο θέσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και το μέλλον της πολιτικής συνοχής που μας έχετε δώσει. Και επίσης θα περιοριστώ σε λίγα με λίγα λόγια να συσχετίσω την ευρωπαϊκή πολιτική με άλλες πολιτικές τις οποίες έχω παρακολουθήσει σε επίπεδο παγκόσμιο, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην Κίνα, τις οποίες είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την περιφερειακή πολιτική, που στηρίζεται στην καινοτομία, και θα δώσω βέβαια και κάποια ε, γρήγορα παραδείγματα. Τα 23 σημεία λοιπόν της εκθεσής σας με οδηγούν ε, σε ιδιαίτερη διατύπωση παρατηρήσεων για 7 θέματα που με ενδιαφέρουν περισσότερο και που μπορούν πιστεύω να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία ανάπτυξη των περιφερειών μας. Καταρχάς λοιπόν και σε δύο χρόνους για να απαντήσουμε στην πολιτική συνοχή ως προς την ποικιλία των ε, περιφερειών, σημαντική πηγή πλούτου που δεν θα πρέπει να ανατρέπεται από την πολιτική συνοχή και ανάπτυξη για την ανα... Ε, έρευνα για την ανάπτυξη και ρόλο της έρευνας και της ανάπτυξης για την ανάπτυξη των ε, περιφερειών και τρίτον θα μιλήσω για τους πιθανούς προσανατολισμούς σε σχέση με την πολιτική phasing in, phasing out, όπου ίσως σήμερα να φαίνεται προφανές ε, το ότι δημιουργούνται ή μπορεί να δημιουργηθούν νέες περιφέρειες. Για το πρώτο σημείο λοιπόν πολιτικής συνοχής, εδαφική συνοχή και η σχέση με την πολυμορφία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι πολιτική συνοχής δεν σημαίνει απαραίτητα μία και μόνη πολιτική ανάπτυξη. Δεν σημαίνει απαραίτητα ανατροπή του πλούτου που μπορεί να προσφέρει κάθε περιφέρεια, ακόμη και οι πιο καθυστερημένες προς την ανάπτυξη, αυτές που ονομάζουμε lagging behind. Επίσης υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθούν όλες οι συνεργατικές δυνατότητες μεταξύ πολιτικής συνοχής και τομεακών πολιτικών που αναπτύσσονται ε, σε οριζόντιο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης τρίτον θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη οι συσχετισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν, οι δεσμοί που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των κέντρων υπεροχής, αριστείας και των πιο καθυστερημένων περιοχικών με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο μέσω του ίντερνετ, παραδείγματι, που επιτρέπει το, την ε, συνεργασία μεταξύ καθυστερημένων και προηγμένων περιφερειών έτσι ώστε και να υποφεληθούν οι μεν των δυνατοτήτων των δε, αλλά και να διερευνηθεί η λόγια των καθυστερήσεων και να προαχθεί η ταχύτερη ανάπτυξή τους. Α, και για το σημείο αυτό επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ήθιστε η Κίνα να θεωρείται χώρα μόνο λυθική χώρα που έχει ε, δυνατότητες εξαγωγικές μόνο χάρη στις χαμηλού κόστους βιομηχανίας της. Όμως τώρα υπάρχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών, των επαρχιών καλύτερα της χώρας και των διαφόρων πόλεων και με πολύ ε, έκπληξη παρατήρησα διαφορές ανάπτυξης που προήχθησαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση και τις επανέλαβε η Κίνα, μάλιστα χορηγώντας και μια σχετική αυτονομία στις επαρχίες, ικανή να προαγάγει την ανάπτυξή τους και να τους επιτρέπει να σχεδιάσουν ε, γραμμές και προσανατολισμούς ανάπτυξης ποικίλε και ε, διαφοροποιημένε. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην σημασία της πολιτικής της ε, καινοτομίας και την, τον αντίκτυπο αυτής στην εδαφική ανάπτυξη και επίσης να αναφερθώ στους στόχους κλειδιά της ανάπτυξης στις περιοχές αυτές υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες για την ε, υλοποίηση μιας στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το 2020 δηλαδή. Έτσι λοιπόν, Στη συνέχεια θα μιλήσω για τα μέσα τα οποία μπορούν να βέλτιστοποιήσουν την πολιτική συνοχής με κυρίως ε, μια στρατηγική phasing in, phasing out και με την ε, παρουσίαση νέων ομάδων περιφερειών όπου πιστεύω ότι χρήσιμο θα ήταν να ε, σχεδιαστεί μια ομάδα περιφερειών αναδυόμενων, θα λέγαμε, ως προς την περιφερειακή καινοτομία. Δύο τέτοια παραδείγματα. Έχουμε από δύο γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφενός μια πρωτοβουλία της μονάδας για τη Γαλλία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για την εκτίμηση των περιφερειακών πολιτικών των 26 ε, γαλλικών περιφερειών, περιφερειών της Γαλλίας, ως προς την περιφερειακή στρατηγική για την καινοτομία, ενδιαφέρουσες προτάσεις και που επιτρέπουν πιστεύω να προσμετρήσουμε την πολιτική που αναπτύσσεται σε περιφερειακό, που καταρτίζεται σε περιφερειακό επίπεδο για την ενίσχυση της περιφέρειας μέσω της καινοτομίας, μέσω της πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης. Δεύτερο παράδειγμα από την Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις, όπου προτείνεται ένα πρόγραμμα top-up scheme ονομάζεται, το οποίο συνδυάζει τις συνεργατικές σχέσεις της κατακόρυφες, σε, από το ευρωπαϊκό στο εθνικό, το τοπικό, το περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση της ανάπτυξης βέβαια και στη συνέχεια οριζόντιες εγκάρσιες σχέσεις ε, συνεργασίας μεταξύ δηλαδή των διαφορών γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή Γενικής Διεύθυνσης για τις Περιφέρειες που αξιοποιεί τα διευθυντικά ταμεία, αλλά και Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις, όπως και τη Γενική Διεύθυνση για την έρευνα που περισσότερο ασχολούνται με την προαγωγή των περιφερειών χάρη στην καινοτομία. Και σε αυτά, με αυτά τελειώνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρουσό. Μας έχει μείνει ένα τέταρτο περίπου για τη συζήτηση. Um, θα ήθελα να σας ενημερώσω, συνάδελφοι, ότι και στην ομάδα εργασία για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας. Αλλά αν έχετε ήδη κάποιες απορίες μπορείτε να τις θέσετε. Ο κύριος Κούρσκι μάλιστα ζήτησε ήδη το λόγο. Οπότε τον έχετε κύριε Κούρσκι. Czy mnie σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονές μας για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν. Ένα τμήμα των παρουσιάσεων το άκουσα προσωπικά με τις παρουσίες στην και ένα τμήμα από το web stream. Ως ε, Πολωνός Ευρωβουλευτής ε, στην παρθενική μου κοινοβουλευτική θητεία δεν μπορώ να μην ε, απηχήσω τις ανησυχίες κάποιων εμπειρογνωμόνων ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προτεραιότητες της ε, ήταν η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι οι χώρες που για πολλά χρόνια βρέθηκαν πίσω από το σιδηρού δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν φυσιολογικά δεν μπόρεσαν να υποφεληθούν ε, από το σχέδιο Μάρσαλ. Οπότε η προτεραιότητα της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης είναι πολύ επίβολο στόχος και πολύ αγαθή πρόθεση. Ακούγεται πολύ ωραία, αλλά είναι ουσιαστικά σαν να παίρνουμε από τη μία τσέπη και να βάζουμε την άλλη. Είναι σαν να παίζουμε το παιχνίδι των παλιών χωρών που είναι και πιο ανεπτυγμένε και μπορούν να επενδύσουν στην καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη ε, αυξάνοντα ακόμη περισσότερο την απόσταση μεταξύ των ε, παλιών χωρών που ήταν ούτω ή άλλω ανεπτυγμένε και των νέων χωρών που είχαν υστερήσει εξαιτία ε, τη παραμονή του διερού παραπέτασμα για πολλά χρόνια. Ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο μας παρουσίασε τώρα τη στρατηγική του 2020 και είπε ότι θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην ευρηματικότητα εις βάρος των ε, προγραμμάτων συνοχής που ενίσχυσαν τη σύγκληση. Νομίζω ότι η σύγκληση είναι πολύ πιο σημαντική γιατί υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και με τη συνοχή και τη σύγκληση θα βελτιώσουμε και την απασχόληση. Είχαμε ήδη τις πρώτες εκθέσεις ε, για τη συνοχή που δείχνουν ότι δυστυχώς ε, επιτείνονται οι διαφορές ε, μεταξύ των περιφερειών στις 27 χώρες μέλη. Κάτι που ίσως δημιουργήσει ε, σε εδαφική διαφοροποίηση, σε περιφέρειες δεύτερης κατηγορίας, κάτι που θα επιδεινώσει την γενικότερη ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη για τις νέες χώρες ε, που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν το δυναμικό που θα μπορούσε κατάλληλα αξιοποιημένο να ωφελήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενιαία αγορά. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στις υποδομές, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και για να εξισώσουμε τις διαφορές αυτές μεταξύ των ε, διαφόρων περιφερειών θα πρέπει να κρατήσουμε πρώτα απ' όλα τους στόχους της συνοχής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ μια ενιαία και ελαστική πολιτική συνοχή. και πιστεύουμε ότι θα πρέπει η παρέμβαση να αντιμετωπίσει τι δημογραφικέ προκλήσει, την παγκοσμιοποίηση, τη φτώχιση κάποιων στρωμάτων του πληθυσμού και να εξασφαλίσει και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Και η περιφερειακή πολιτική είναι σημαντικό εργαλείο και τη ε, πολιτική συνοχή για να εξασφαλίσουμε και την οικονομική και την κοινωνική συνοχή γιατί δεν θα πρέπει ε, ε, παρά τη θέλησή μας να δημιουργηθεί ένα νέο σιδηρού παραπέτασμα εξαιτία των οικονομικών και κοινωνικών διαφορών. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να καλύψουμε αυτά τα κενά και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των παλιών και των νέων χωρών και θα πρέπει σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα βήμα πρόοδου και να επικεντρωθεί αφού καλύψει αυτές τις διαφορές στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία. Βέβαια, σήμερα κάτι τέτοιο θα ήταν πρόωρο και πολύ πρόημο και θα οδηγούσε σε ένα de facto νέο σύνδρομο της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Γι' αυτό και είμαστε αποφασιστικά και κατηγορηματικά ως ευρωβουλευτές νέων χωρών υπέρ της διατήρησης Τη συνοχή ως προτεραιότητα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε παρόμοιες ευκαιρίες και στις δύο πλευρές Ευρώπης για χώρες που για πολλά χρόνια δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν φυσιολογικά. Σας ευχαριστώ κύριε Κούρσκι. Το λόγο έχει ο κύριος Βανίστεροι. Ευχαριστώ. Το κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε αλλαγές ή όχι, αν είναι νωρίς ή όχι, μα τώρα μιλάμε για την περίοδο 2013-2020 για νέα πολιτική συνοχής. Οπότε δεν ξέρω γιατί λέτε αν είναι νωρί ή αργά. Τώρα μιλάμε για τη νέα αρχιτεκτονική. Στη νέα συνθήκη αναφέρεται η περιφερειακή διάσταση, η περιφερειακή συνοχή και αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι μήπως υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος για να πετύχουμε την ισορροπία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κάθε χώρα. Το μέσον υπάρχει στην πράσινη βίβλο. Ακούω να λέτε ότι η εδαφική συνοχή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία γεωγραφικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συγκέντρωση και από την άλλη μεριά να έχουμε συνεργασία. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το εξή. Άκουσα τον τελευταίο κυρίως ομιλητή να αναφέρεται σε νέα μοντέλα ώστε να πετύχουμε θέμενη αξία ακόμα περισσότερη και οι διάφορες γενικές διευθύνσεις αναπτύσσουν νέες ιδέες. Τώρα, για τα αυτά που συμφωνούμε με τις χώρες. Κοιτάξτε, μια περιφέρεια η οποία δεν έχει όραμα για την ανάπτυξη και δεν καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις. υπεθρός, οτιδήποτε. Ή σε σχέση με νέες ε, πρωτοβουλίες, έρευνα και ανάπτυξη. Ε, όχι διότι θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για να συμμετέχει μια περιφέρεια. Αν δεν μπορεί, όχι. Αυτοί όμως που μπορούν και θέλουν και έχουν όραμα, εν μάλιστα και της στρατηγικής 2020 που μιλάει για πιο ευθύ και αηφόρο και πράσινη ανάπτυξη, ναι, να συμμετέχουν. Αν το βρίσκουν πολύ δύσκολο, ας μην το κάνουν, ας μην συμμετέχουν. Για μένα αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Σεν Κέλλη. Δύο λόγια μόνο για διευκρίνηση. Τα στοιχεία που δίνονται για τις περιφέρειες Ευρώπης, 55% νομίζω βρίσκονται κάτω από το 75% επί του μέσου άρου του ΑΕΠ, 30% πάνω, 15% ε, πάνω. Ποια είναι ακριβώς τα στοιχεία, ποιες είναι οι αναλογίες, σε τι αναφέρονται και γεωγραφικά αυτές τις περιοχές που εντοπίζονται. Το άνω 15% είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης, το άνω 30% και το καθεξής. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσει. Κονδύλια επίσης τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί από μια περιφέρεια δεν θα πρέπει να πηγαίνουν ε, σε ένα κράτος, αυτό μας είπατε αν κατάλαβα καλά, δηλαδή να ε, επανέρχονται στον εθνικό προϋπολογισμό για να χρησιμοποιηθούν σε άλλα σχέδια. Μήπως όμως έτσι ε, οθήσουμε τα κράτη να υπερβάλλουν και να λένε «Α, τόσα πολλά κονδύλια που δεν αξιοποιήθηκαν τα ξαναπαίρνω εγώ και τα ξανααξιοποιώ». Παρακαλώ, κύριο Σόλεσνακ. Νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι μιλούμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής σε ευρύς όρους τώρα, αλλά όχι μόνο με προοπτική την Ευρώπη του 2020, αλλά και αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή το συντονισμό περισσότερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν υπάρχουν κάποιες ατέλειες, ασφαλώς και αυτές απορρέουν από τα όσα μας αναφέρατε τώρα τα οποία βρίσκω πράγματι πολύ χρήσιμα, τροφή για σκέψη. Αλλά θα ήθελα να πω και στα όσα είπε ο κύριο Κούρσκι ότι βεβαίω έχουμε κάποια προβλήματα ω προ τι υποδομέ. Εμεί τα νέα κράτη, τα κράτη που πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε προβλήματα ω προ του δρόμου αλλά και άλλε υποδομέ. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση και ακόμα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κάλυψη του χαμένου εδάφου. Όταν μιλούμε λοιπόν για 2013 ή για 2020, ασφαλώ δεν μπορούμε να ε, περιμένουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες μας τις, προσπά... μας τις προσπάθειες μέχρι τότε. Απλώς θα έχουμε πάρει μια κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι πρέπει τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να μεριμνήσουν έτσι ώστε να έρθει η ώρα για τις υποδομές στην προσεχή περίοδο να είναι έτοιμες να λάβουν πιο δραστήρια δράση. Βεβαίως και υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις, ουσιώδεις προκλήσεις, πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει επανελειμμένα εδώ στην διεθνή ή παγκόσμια ανταγωνιστική σχέση που έχουμε, όχι μόνο με την Κίνα, αλλά και με άλλες αναδυόμενες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για εκπαίδευση, πρέπει να μιλήσουμε για κατάρτιση, για νέες και καθαρές τεχνολογίες. Η Πολωνία είναι ένα παράδειγμα για το οποίο έχω ανησυχίε, διότι υπάρχουν ορισμένοι τομεί του οποίου βλέπω να καθυστερούμε τόσο που θα ξεκινήσουμε τι προσπάθειε όταν θα είναι πιο, πια πολύ αργά. Και στι ταπάνε για τι νέε τεχνολογίε και στι ταπάνε για την εκπαίδευση. Ε, εάν δεν πάρουμε, τουλάχιστον εμεί στην Πολωνία, ε, άμεσα τώρα, ε, αμέσως ε, κονδύλια, θα είναι πολύ αργά πια για να καλύψουμε το χαμένο έδαφο. Και για τον κύριο Σλάχτερ θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό κρίνεται την καθυστέρηση, πώς ακριβώς κρίνεται και εξολογείται την καθυστέρηση μεταξύ κρατών μελών και χωρίς βέβαια να θέλω να μιλάω για παλαιά ή νέα κράτη-μέλη, θα ήθελα να γνωρίζω τι διαφορές βλέπετε και πού μας τοποθετείτε εμά για την δημοσιονομική στήριξη, την οικονομική στήριξη, πού είναι τα κενά και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαλεμένο έδαφος και στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα τις καθαρές τεχνολογίες. Δυστυχώς ξέρω την απάντηση. Έχουμε φοβερά κενά και λήψεις στις υποδομές. Και πολλά θα πρέπει να κάνουμε για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Οπότε και στην έρευνα και στην τεχνολογία και στην καινοτομία υπάρχει τεράστια ε, αδυναμία αυτό το χώρο, τεράστια υστέρηση. Εγώ Ακριβώ επειδή έχουμε αυτή την υστέρηση, πιστεύω ότι θα πρέπει ακριβώ να επενδύσουμε στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη. Οπότε διαφωνώ ριζικά με αυτά που είπε ο συνάδελφο Κούρσκι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένα έχει τη δική του γνώμη. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στου εμπειρογνώμονε για να σχολιάσουν ό,τι θέλουν από αυτά που ακούσαμε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να εμείνω σε κανένα δύο σχόλια που έγιναν. Συμφωνώ με τον κύριο Κούρσκι σε ό,τι αφορά την έμφαση στην καινοτομία και τη σχέση με τη στρατηγική του 2020. Υπάρχει ένας κίνδυνος, αν υιοθετηθεί μια προσέγγιση από, τα, από την κορυφή προς τη βάση, να υποβαθμιστούν κάποιες αναπτυξιακές προτεραιότητες, ε, κυρίως των ε, λιγότερων ανεπτυγμένων περιφερειών. Και αυτό υπογραμμίστηκε στην έκθεση Μπάρκ που πρότεινε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την έμφαση που δίνεται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετικές περιοχές και περιφέρειες. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του Λάμπερτ Βανίστερόι, η προσέγγιση της εδαφικής συνοχής δίνει νέα πρίσματα και νέες προοπτικές ό,τι αφορά την ελαστικότητα ή την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα σε εδαφικό επίπεδο. Είδαμε κάποιες προ... πρωτοβουλίες για τις μακροπεριφέρειες, για τα δίκτυα και διάφορες πλατφόρμες διαπεριφερειακής συνεργασίας ή κάποιες τοπικές πρωτοβουλίες όπως το Urban και το Leader. Επίσης, βλέπουμε τι συμβαίνει στι εθνικές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, για παράδειγμα. Πάντως, ε, μπορούμε να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τέτοιου είδους προσέγγιση και όπως ε, αναφέρθηκε στο παρελθόν, τέτοιου είδους ε, προσεγγίσεις είναι καλύτερο να γίνονται από την, από την βάση προς την κορφή και όχι αντίστροφα. Σε ό,τι αφορά την μεταφορά κονδυλίων ή τη χρήση τους σε άλλες περιοχές, όντως υπάρχει κίνδυνος κυρία Κέλλη και είχαμε τέτοια εμπειρία για, ένα, ε, για μια πρόταση, για ένα αποθεματικό σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και εκεί χρησιμοποιούνταν κονδύλια από περιοχές που, που δεν είχαν εντυπωσιακέ επιδόσεις ή που υποχρησιμοποιούσαν τα κονδύλια τους σε περιφέρειες που είχαν καλύτερο βαθμό επιδόσεων. Ο κύριος Λέγκ, παρακαλώ, σε πέντε λεπτά θα σταματήσει η διερμηνία, οπότε να είστε συνοπτικοί. Ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας ρωτάτε. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Την ε, εδαφική συνοχή πρέπει να τη δούμε σαν ένα παράθυρο ευκαιριών, γιατί μπορούμε να βάλουμε στην πολιτική καινούριο αέρα. Είναι προς όφελός μας. Θέτοντας εφαρμογή την πολιτική συνοχή, μπορούμε επίσης να σκεφτούμε και άλλη διάσταση της συνοχής που δεν υπάρχει στη στιγμή που είναι ε, πολιτιστική και άλλες. Δεύτερο σχόλιο. Πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα να γίνει γκέτο για τους φτωχούς η πολιτική συνοχής. Και γι' αυτό και πρέπει να πάμε προς μια νέα κατεύθυνση. Πολύ σοβαρή κριτική για την πολιτική συνοχής εντοπίζει τρεις χώρους όπου είναι σημαντική και αναγκαία η πολιτική συνοχής. Παραδοσιακές υποδομές, γιατί υπάρχουν απομονωμένες περιφέρειες βέβαια, πολύ φτωχές περιφέρειες, ιδιαίτερα φτωχές, και τρίτον διασυνοριακή συνεργασία. Γιατί είναι αδύνατο να βρούμε μια καλύτερη θέση. Μην μπούμε στην παγίδα. Ένα άλλο σχόλιο ο Ζαν σίγουρα έχει να πει περισσότερο. Όταν μιλάμε για την συνοχή, σε επίπεδο χωρών είμαστε επιτυχείς. Οι κυβερνήσεις είναι ευτυχείς με αυτή. Μπράβο. Σε περιφερειακό επίπεδο οι καλές στατιστικές μπορούν να κάνουν κόλπα και να πούνε ότι ναι ή όχι. Αλλά οι διαφορές είναι μικρές. Και μέσα στις χώρες παρατηρούμε μεγάλες διαφορές στην ανάπτυξη. Και αυτό είναι το ζήτημα. Είναι το δικό μας πρόβλημα αυτό ή όχι. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για τον κάθε ομιλητή. Παρακαλώ. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις περιφέρειες... Είμαι... Βάσει τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, δεν είναι δική μου επινόηση, ε, περιφέρειες που βρίσκονται κάτω από το 75% του κοινοτικού ΑΕΠ είναι 68 στις 27 χώρες μέλη και 20 στις 15 και στις 48. Οπότε 28 και 40 μας κάνει το 68. 67 περιοχές του ΝΑΤΣ 2, δηλαδή 80% στην Ευρώπη των 15, 4% στην Ευρώπη των 12. Δηλαδή 81 περιφέρειες από 271, δηλαδή 30% των περιφερειών ε, μεταξύ 60 και 100 και οι υπόλοιπε μεταξύ 100 και 150. Δηλαδή 97% στις παλιές ε, χώρες ε, μέλη και 75%. 100 στις νέες. Δηλαδή 104 από τις 271 περιοχές βρίσκονται σε πολύ μέτρια κατάσταση. Ο κύριος Ρουσό. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά την ανάγκη της διασυνοριακής συνεργασίας που αφήνει κατά μέρους όλες τις ε, περιφέρειες τις εσωτερικές. Και ίσως καλύτερα να μιλήσουμε για διακρατική συνεργασία και όχι διασυνοριακή. Θα ήθελα να φτάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσης διάταξης πριν να ευχαριστήσω τους εμπειρογνωμονές μας, να ενημερώσω τους συναδέλφους για τις χθεσινές αποφάσεις των συντονιστών. Καταρχήν, ε, την έκθεση ε, για τη Μαδέρα και τις Αζόρες ε, θα την αναλάβει και πάλι η Προεδρία, η Πρόεδρος η έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, την γνωμοδότηση την ε, ανέλαβαν οι φιλελεύθεροι και την, το θέμα της απλούστευσης ε, του ερευνητικού προγράμματος, το ΕΛΚ. Επίσης, ε, οι συντονιστές πρότειναν να ληφθεί απόφαση μέχρι τη Δευτέρα 6 το απόγευμα, το αργότερο, για το κατά πόσο θα ζητηθεί έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής που θα αποτελέσει τη βάση για την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Επίσης συμφωνήσαμε 7, έξι μάλλον ε, εκθέσεις και μία έκθεση εφαρμογής. Η έκθεση εφαρμογής αφορά την ε, στρατηγική έκθεση του 2010, θα την αναλάβει το ΕΛΚ και η έκθεση για το στόχο 3 επίση είναι του ΕΛΚ. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες ανέλαβαν την έκθεση για τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ταμείων. Τις δημογραφικές αλλαγές ε, θα τις αναλάβουν στην έκθεσή τους πάλι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Για τα προβλήματα απορρόφησης ε, θα συντάξουν έκθεση φιλελεύθεροι. και οι μεταρρυθμιστές συντηρητικοί θα αναλάβουν την έκθεση για τις αστικές περιφέρειες. Ενώ οι, οι πράσινοι επίσης αναλάβουν μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη για το, για το θέμα. Θα σας στείλουμε πιο ακριβείς πληροφορίες για τους συγκεκριμένους τίτλους των εκθέσεων ίδιας πρωτοβουλίας. Επίσης το θέμα των μηχανισμών κυρώσεως θα, τα, θα το συζητήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση όπως πρότεινε η Άλντε. ό,τι αφορά το Συμβούλιο του Τολέδο την απόφαση σχετικά θα την ε, λάβουμε στην επόμενη μας συνεδρίαση του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ καρποφόρη συζήτηση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες που θα έχουμε τη χαρά να δούμε και αργότερα στην ομάδα εργασίας. Σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση.